Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τις, τη συνεδρίασή μας και να σας καταρχάς για τις αποφάσεις της συνεδρίασης των συντονιστών. Συνεδρίαση που είχαμε χθε το απόγευμα. Εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, ως προς αυτό αποφασίσαμε ότι θα περιμένουμε μερικές μέρες ακόμα προκειμένου να γίνουν κάποιες ε, προτάσεις και από τις ε, πολιτικές εκείνες ομάδες που δεν έχουν υποβάλει γραπτές προτάσεις ακόμα. Όσον αφορά τις αντιπροσωπείες επιτροπής μας αποφασίσαμε δύο μερομηνίε. Κορσική και Σαρδινία, καθώς επίσης και Σουηδία, εβδομάδα 25 και εβδομάδα 29. Δεν προβλέπονται όμως ημερομηνίες για την επίσκεψη στο Βερολίνο και στη Βουλγαρία ακόμα και περιμένουμε από τις πολιτικές ομάδες και ιδίω από το ΕΛΚ και τους αλιστές να καταφέρουν να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατό γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ενημερώσω και την διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, το συντομότερο δυνατό όσον αφορά την Regional State Day. Μιλώντας και με τον Επίτροπο Αλμούνια, είπαμε ότι θα τον προσκαλέσουμε και αυτόν και τον Επίτροπο Χάν στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει το Φεβρουάριο, προκειμένου να του εξηγήσουμε τις ε, προτάσεις ε, της Επιτροπής μας για την ημέρα υποστήριξης προς τις περιφέρειες. Προτείναμε να συνεδριάσουμε κατά τη διάρκεια της ημερομηνίας προβλέπεται για την Επιτροπή μας. Αν δεν γίνει δεκτή η ημερομηνία αυτή, τότε θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να έχουμε τον κύριο Μάτιν από την DG Radio και τον κύριο Κόπμαν για, τη δύο αυτήν υπεύθυνη για την ημέρα αυτή. Επίσης θα προτιμάσουμε τις προφορικές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένω επίσης να συμβάλλετε κι εσείς ε, από τις πολιτικές σας ομάδες για τη σύνταξη των προφορικών αυτών ερωτήσεων. Όσες πολιτικές ομάδες βέβαια ενδιαφέρονται. Επίσης, ε, αποφασίσαμε και για πρωτοβουλία που προέρχεται από το ΕΛΚ όσον αφορά την ε, περιοχή των Άλπαιων. Προβλέπετε για το ζήτημα αυτό μια προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και περιμένουμε όμως και πάλι συγκεκριμένες προτάσεις από τις πολιτικές ομάδες που θα έρθουν επιπλέον στα όσα έχει ήδη υποβάλει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτές είναι οι αποφάσεις των συντονιστών και στο τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης αυτές θα εγκριθούν επισήμως. Ας περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημέρησιας διάταξης. για Ολμπρίχτ, ενημέρωση σχετικά με τις ε, ενεξελίξει διοργανικές διαπραγματεύσεις για την έκθεση για την οποία είναι υπεύθυνο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δεν έχουμε ακόμα μαζί μας τους σκιώδεις εισηγητές. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο. Γιάννη, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να πάρεις το λόγο να μας παρουσιάσει την κατάσταση. So you can come here. Could somebody activate the mics? Μπορεί κάποιος να βάλει μπρος τα μικρόφωνα. In, in case you are, it's working here. Εδώ πάντως δουλεύει το, το μικρόφωνο. Μ' ακούτε? Ωραία, μ' ακούτε. Εντάξει, τώρα λειτουργεί. Λοιπόν, πολύ καλά. Μπορώ να σας ενημερώσω σε σχέση με το πώς διαμορφώθηκαν τα πράγματα στον τριμερή διάλογο και τι συνέβη σχετικά. Νομίζω είναι πραγματικά σημαντικό κάποια στοιχεία για το ΕΦΤΕ να ληφθούν υπόψη που όσον αφορά τον βασικό κανονισμό πρέπει να αποσαφινιστούν διότι επηρεάζονται σε σχέση με αυτόν. Υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με την Συμφωνία εταιρική Σχέσης. Ένα σημείο επί της ουσίας ε, σε σχέση με τη συνθήκη αφορά τις πτυχές ε, των πόλεων, δηλαδή την αηφορία και τη βιωσιμότητα όσον αφορά τα κέντρα, τα αστικά κέντρα της πόλης στο αρχικό κείμενο αναφερόντουσαν οι πόλεις που προτείνονται από τα κράτη-μέλη για τέτοιες ε, δράσεις για την αηφορία. Αυτό το τμήμα μετά την πρότασή μας τροποποιήθηκε όμως. Και έτσι <clears throat> δεν αποτελεί μέρος ε, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Τουλάχιστον όχι ο κατάλογος αυτών των πόλεων που κανονισμούς και κριτήρια υλοποιούν προς μια τέτοια αηφορία, αηφόρο δράση. Με άλλα λόγια, οι διατάξεις και οι κανονισμοί για μελλοντικούς τέτοιους πίνακες και την ένταξη σε αυτούς πόλεων για την αηφορία. Στον βασικό λοιπόν κανονισμό άλλαξε αυτό και γι' αυτό στον τριμερή διάλογο ακολουθήσαμε αυτή την απόφαση, αυτό ε, μπόρεσε να γίνει, υπό την προσπάθεια προσδιορισμού, ορισμού των πόλεων. Να σας υπενθυμίσω ότι αρχικά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης ε, προέβλεπε για τέτοιου είδους φόρες δράσης. και στον δικό μας τριμερή διάλογο προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε και να δούμε ποιο είναι το νόημα αυτών των 5% ποσοστού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες να περιγραφεί και να διαπιστωθεί το Πρώτον, ε, τα μέτρα τα οποία μπορούν να επικεντρώνονται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δράση και δεύτερον τα κράτη-μέλη να πιστούν και να κινητοποιηθούν λειτουργούσε τέτοιε περιφέρειες ή περιοχές να ταυτοποιήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά είχε υπόψη μόνο πόλεις ή αστικά κέντρα. Εμείς θέλουμε να έχουμε την δυνατότητα να υπάρξει κατάρτιση ενός επταετούς ε, ε, σχεδίου. Και δεύτερον, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και για την Επιτροπή και για μας. Επιθυμούμε οι αρχές στις πόλεις αυτές, δημοτικά συμβούλια, δήμαρχοι, να έχουν την δυνατότητα μέσα στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων να δρουν διατηρώντα την αρμοδιότητα ανάληψη πρωτοβουλία και δράση. Να υπενθυμίσω ότι σε σχέση με τι πόλει και τι εταιρικέ σχέσει, τα κριτήρια και οι διατάξει καθορίζονται για τις πόλεις και καθορίζεται και ένα 5% ποσοστό από το ΕΤΠΑ για αυτές και η μεθοδολογία για τον στόχο αυτό του 5% καθορίζεται. Τώρα, όσον αφορά αυτή τη μεθοδολογία, η μέθοδο, τι γίνεται. Δια, διατυπώνεται το περιβόητο ερώτημα των ITIs. Είναι δεσμευτικού χαρακτήρα τα ITIs μέσα στο πλαίσιο του 5% αυτού του ποσοστού. Του του λεχθέντος τώρα η επιλογή ή όχι, να το πω καλύτερα, οι δημοτικές αρχές μπορούν με ε, θελοντικό ε, χαρακτήρα να μπορέσουν να αποφασίσουν αν ε, θα ακολουθηθεί ένα τέτοιο ITI ή όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το 5% για τις πόλεις. Η μεθοδολογία θα πρέπει να καθοριστεί και στο τέλος, τέλος και αυτό σε σχέση με την ομάδα εργασίας και στον τριμερή διάλογο έχει προχωρήσει. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό λοιπόν από πλευράς μας να αποσαφινιστεί το πρόβλημα της αντιπροσωπείας, το θέμα τι θα γίνεται με τις αντιπροσωπείες. Θεωρούμε ότι αυτό το οποίο δημιουργεί την πρόσθετη, πρόσθετη αξία στο τέλος είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στις περιφερειακές και τοπικές αρχές και η άσκηση πρωτοβουλίας από εκείνες, διότι αυτή η μετάθεση, η μεταφορά αρμοδιότητας ε, ευθύνη μπορεί να επηρεάσει τα σχέδια και τις εξελίξεις ε, όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση. Όμως η άλλη πλευρά δεν είναι πρόθυμη να επιτρέψει να δεχθεί αυτή την μετάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών αντιμετωπίζουμε, βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε αυτό το πρόβλημα. Το γενικότερο ζήτημα είναι αν διατηρηθεί αυτό το 5% θα πρέπει να μπορεί να απορρέει πρόσθετη αξία ως αποτέλεσμα από αυτήν. Διότι αν δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα νέων σχεδίων με πρόσθετη αξία τότε δεν έχει νόημα αυτό το 5% ως ποσοστό πρέπει να δράσει ώστε από κοινού κοινά μέτρα και δράσεις σε σχέση με τους πολίτες επιτόπου να μπορούν να αναπτυχθούν. Ένα action urban για παράδειγμα, κάτι παρόμοιο όπως την δράση για τις πόλεις με διαφορετικό χαρακτήρα αλλά κάτι παρόμοιο. 5% λοιπόν για τις ε, περιοχές των πόλεων. Αυτό επιθυμούμε. Τώρα αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου και αναμένουμε και την απόφαση για τις αρμοδιότητες. Ποιος θα έχει την τελική αρμοδιότητα. Πάλι από πλευρά του Συμβουλίου αυτή η απόφαση. Υπήρξαν και κάποια κάποιες τριβές, κάποιες ε, αντιρρήσεις, όχι τόσο από το Συμβούλιο, αλλά από τους περιφερειακούς εταίρους, όσον αφορά μια πλατφόρμα, όσον αφορά δηλαδή μια κοινή βάση πόλεων. Υπάρχουν πόλεις που στο πρόγραμμα της καινοτόμου δράσης θέλουν να συμμετάσχουν, όμως τα Δημοτικά Συμβούλια ισχυρίζονται, οι σύμβουλοι, ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναγκαιότητα για μια νέα τέτοια πλατφόρμα. Εμείς υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζουμε ότι μια τέτοια πλατφόρμα μπορεί να συνεισφέρει στην διάχυση διάδοση γνώσεων και ανταλλαγή βέλτιστων εμπειριών. Και νομίζουμε ότι μέσα στο πλαίσιο αυτού του ποσοστού πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή τη δράση, διότι διαφορετικά είναι δύσκολο να υπάρχει διαδραστικό διαδραστικός χαρακτήρας, αμφίδρομη δράση, feedback. Κατά τα άλλα, Ω ένα είδου πιλωτικό σχέδιο μπορεί κάτι να λειτουργήσει. Χωρί μια πλατφόρμα τέτοια δεν μπορεί κανεί να γνωρίζει αν παράγεται πρόσθετη αξία ή όχι. Εμεί είμαστε υπέρ της διατήρησης, της διαφύλαξης αυτής της αστικής πλατφόρμας των πόλεων, αλλά μόνο με το 5% και με τις καινοτόμε δράσεις φυσικά από κοινού προτείνει 5,5% ε, του ΕΠΑ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις ε, Υποστηρίξαμε αυτή την πρόταση. Αυτό το ποσοστό θα προβλέπεται για τα μίνι προγράμματα σε σχέση με τις πόλεις. Υπάρχει έτσι αυτή η δυνατότητα μέσω του 0,2 διορθώνει ο εισηγητής 0,2% να ξεκινήσουν και να μπορέσουν να λειτουργήσουν σχέδια που θα έχουν κάποιο ε, πρόσθετη αξία. Όπως προανέφερα στα άρθρα 7 και 8 έγκυνται τα κυριότερα προβλήματα για την αντιπροσωπεία, την μεταφορά, μετάθεση ε, αρμοδιοτήτων. Υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο το οποίο συζητήσαμε αλλά δεν το ολοκληρώσαμε, δεν καταλήξαμε σε απόφαση. Υπήρξε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες δηλαδή το, από πλευράς επενδύσεων. Αυτό ήταν το θέμα που συζητήσαμε. Θεματολογικά οι στόχοι είναι κάτι που στον βασικό κανονισμό περιγράφονται ήδη. Δεν καθορίζουμε, δεν προσδιορίζουμε εμείς εκ νέου αυτούς τους στόχους. Εκείνο το οποίο όμως είναι ένα νέο καινούριο στοιχείο είναι η θεματολογική επικέντρωση ε, θεματολογική εστίαση τι θα γίνει στις λιγότερο, για παράδειγμα, ανεπτυγμένες ε, ε, περιφέρειες, στις ήμι ανεπτυγμένες περιφέρειες και εκείνες ε, για τις οποίες προβλέπεται αυτή η θεματική, θεματολογική εστίαση. Το Συμβούλιο θεώρησε ότι αυτό το σημείο μόνο τότε μπορεί να αποσαφινιστεί όταν οι θεματολογικοί στόχοι θα έχουν αποσαφινιστεί σε σχέση με το βασικό κανονισμό. Τώρα τι κάνουμε. Εργαζόμαστε σε σχέση με την δρομολόγηση της λειτουργικότητας αυτών αυτών των θεματικών, θεματολογικών στόχων. Πρέπει όμως πρώτα οι προτεραιότητες για τις επενδύσεις να προσδιοριστούν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρέπει να αποσαφινιστεί τι θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει όσον αφορά τις προτεραιότητες σε σχέση με τις επενδύσεις. Δεν γνωρίζω τώρα, Πρόεδρε, τι να κάνω. Να απαριθμίσω τις επιμέρους προτεραιότητες ή όχι. Ίσως θα μπορούσα να δώσω μια περίληψη εν συντομία. Κάποιες από τις προτάσεις μας υποστηρίζονται από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως η πρόταση υπό άλλο πρίσμα θα πρέπει να εξεταστεί και να προσεγγιστεί. Για παράδειγμα, δεν επαρκεί να περνάμε από το ένα σημείο στο άλλο. Δεν επαρκεί. Συμφωνούμε, ναι μεν, αλλά θεωρούμε ότι και κάποια άλλη προσέγγιση θα πρέπει επιπρόσθετα να ληφθεί υπόψη. Διαφοροποίηση. Επί της ουσίας δεν υπάρχουν λοιπόν διαφορές, αλλά μόνο όσον αφορά την προσέγγιση υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις. Η μεγαλύτερη θα έλεγα διαφορά είναι το θέμα της μεταφοράς όσον αφορά την, από το 7 στο 4 και της ε, ε, μείωση των εκπομπών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα, την μείωση δηλαδή των εκπομπών άνθρακα στην, ε, στον, στην ατμόσφαιρα και σε σχέση με την μεταθεσή από το 7 στο 4. Δεν θα ήθελε το Συμβούλιο συνολικά να μετατεθεί το σύνολο της, των μεταφορών από, στο, από το 7 στο 4 αλλά η κινητικότητα τουλάχιστον σε σχέση με τις πόλεις με τα αστικά κέντρα θα έπρεπε να λειτουργήσει έτσι και έτσι συμφωνούμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή εμείς ως προς αυτά. Όσον αφορά τα άλλα στοιχεία καταβάλαμε προσπάθειες ε, ε, και έγινε λόγος και εχθές ε, για την FEE e εξειδίκευση, εξειδίκευση της αγοράς ε, και η δημιουργική βιομηχανική κλάδη που είναι ένα από τα στοιχεία πυρήνες και κλειδιά έχουν ταυτοποιηθεί. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια να μπορέσει το κείμενο να προσαρμοστεί σε σχέση να, λάβει υπόψη αυτά τα στοιχεία. Μόνο οι διαφορές που βρίσκονται. Βρίσκονται μεταξύ της δικής μας θέσης και ε, των άλλων δια... εταίρων στη διαπραγμάτευση. Επειδή το Συμβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ότι ο πίνακας δεν πρέπει να αποτελεί μέρος ε, των προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις και ότι πρόκειται μάλλον για ένα θέμα περισσότερο αρμοδιότητας των πόλεων. Είναι μέρος αυτών των ε, μέτρων οι προτεραιότητες και ο κατάλογος είναι τμήμα αυτών των μέτρων ή όχι ή πρόκειται για κάποιο άλλο πλαίσιο. Τώρα, αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας κατάλογος αυτών των μέτρων. Αν συνέβαινε λοιπόν κάτι τέτοιο, σε περίπτωση που δεχόμαστε εμείς αυτό, τότε θα έπρεπε οι προϋποθέσεις όλης της ε, λίστας, όλου του καταλόγου να υλοποιηθούν και όχι να γίνει κάτι υστερότερα, διότι αυτό θα, ήταν υπερβολικά, ε, θα ερχόταν με υπερβολική καθυστέρηση. Λοιπόν, είτε όλα θα πρέπει σε ένα γενικό πλαίσιο να επιτρέπονται και να μπορούν να λειτουργήσουν ή θα υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο εξειδικευμένη, πιο χειροπιαστή μια απόφαση πρέπει να ληφθεί από μας ως προς αυτό. Αυτή είναι η συζήτηση όπως διαμορφώθηκε. Μπορείτε να θυμηθείτε τι έγινε και με τον χρονορίζοντα και τις στρατηγικές προτεραιότητες για το 2020, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόταση για οριζόντια μέτρα. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει στο προήμιο να ενταχθούν αυτά και να καθορίζονται μέσα στο ίδιο το προήμιο. Διαρωτώμεθα λοιπόν εδώ, αυτά που βρίσκονται στο προήμιο ή στις αιτιολογικές σκέψεις, στα σκεπτικά, έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα ή είναι μόνο εισαγωγικά. Είναι νομίζω κάτι σημαντικό και ορθό αυτό, αλλά πρέπει να πω από την άλλη πλευρά ότι θεωρώ ότι αυτά τα οποία στις προτεραιότητες για τις επενδύσεις καθορίζουμε θα πρέπει να πολύ ισχυρότερα να λαμβάνονται υπόψη και μπορώ κάποια από αυτά τα στοιχεία να σας τα αναφέρω. Η co-generation, συμπαραγωγή, Ουσιαστικά συμφωνούμε για την συμπαραγωγή co-generation, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Πιο συγκεκριμένοι ως προς αυτό. Θα θέλαμε αυτή την πτυχή να την δούμε με το Ταμείο Συνοχής από κοινού, που εκεί θα μπορούσε να ε, εντασσόταν. Τώρα, το ίδιο πρόβλημα από την άλλη πλευρά όπως και με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης θερμότητας, απορρέει και στον τομέα των, ε, ε της στέγασης ε, των διαμερισμάτων, κτηρίων Όλα αυτά είναι υπερβολικά γενικόλογα. Τι θα γίνει, δημόσια κτίρια, δημόσια ε, κρατικής ιδιοκτησίας ή ιδιωτικά διαμερίσματα και κατοικίες. Στα περισσότερα κράτη-μέλη από την κρατική πτυχή, από το τον κρατικό χαρακτήρα αυτών των κτιριων ξεκινά κανεί. Γι' αυτό θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει λόγο για public και private, δηλαδή ε, κρατικά και ιδιωτικά κτίρια. Και έτσι τα ιστορικά κτίρια μπορούν να καλύπτονται. Γιατί τα ιστορικά, θα μπορούσε κανείς να λαμβάνει υπόψη ότι και τα παλαιά και τα νεότερα θα λαμβανόντουσαν, θα καλυπτόντουσαν. Αλλά πρέπει και η αποδοτικότητα της ενέργειας και αυτή να λαμβάνεται υπόψη. Και επειδή θέλουμε στα ιστορικά, ιστορικού χαρακτήρα να μπορούν να αναφέρονται, τότε πρέπει να δούμε γιατί δεν θα μπορούσε αυτό να ενταχθεί στον κανονισμό. Η άλλη πλευρά δεν είναι αναγκαίο να ενταχθεί στον κανονισμό. Καλύπτεται από την οδηγία, λέει, αυτή η πτυχή για την αποδοτικότητα της ε, ε Τη της παραγωγής και χρήσης ενέργειας. Θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα και ε, η βελτίωση, βέλτιστη επίδοση ε, θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη και δεν μπορεί κανείς να επιχειρηματίσει ότι είναι το ίδιο αυτό όσον αφορά για παράδειγμα ιστορικού χαρακτήρα κτίρια ή νέα κτίρια, νέες κατασκευής. Δεν θέλω να επισέλθω υπερβολικά σε λεπτομέρειες τώρα, εντάξει. Θα ήθελα να πω ότι θα προσπαθήσουμε από πλευράς ουσίας να έχουμε το ίδιο περιεχόμενο που θα εντάσσεται στο κείμενο. Και αυτό θέλω να περάσει ως μήνυμα. Δεν προσπαθούμε να, αλλοιώσουμε κάτι, αλλά προσπαθούμε στο τέλος τέλος να δούμε ότι το αποτέλεσμα μπορεί τελικά να μην είναι εκείνο ακριβώς το οποίο θα ήταν αν είχαμε την αποκλειστική εντολή εμείς για τη διαμόρφωση αυτών των πραγμάτων. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε αυτό το περιεχόμενο αυτής της ουσίας και σε σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δίνουμε μάχη για να τα καταφέρουμε. Ούτως έχουν τα πράγματα. Και στις ε, τέλη Ιανουαρίου θα έχουμε μια συνάντηση πάλι για να ξανασυζητήσουμε αυτά τα πράγματα και θα γίνει λόγος εκεί για τις προτεραιότητες επενδύσεων και τους δείκτες. Θα προσπαθήσουμε τους δείκτες να μην τους αφήσουμε στον κανονισμό διότι οι δείκτες που υφίστανται αυτή τη στιγμή συνδέονται πάρα πολύ στενά με τον κανονισμό. Και αυτός ο κατάλογος θα έπρεπε να είναι μέρος μιας κατεκτέλεσης, κατεντολήν πράξης και θεωρώ ότι εμείς ως Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να επεξεργαστούμε τους δείκτες αυτούς. Είναι τεχνικού χαρακτήρα νομικά ιδιαίτερα τεχνικά θέματα. Θα είναι δύσκολο με άλλα λόγια λοιπόν, ας το πω έτσι, να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα και με τα κράτη-μέλη, μια και θέλουν να διατηρήσουν αυτούς τους δείκτες από πλευρά τους. Κατά τα άλλα η ατμόσφαιρα ήταν και είναι θετική, συνεργαζόμαστε με επικοδομητικό πνεύμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε, να διευκρινίσουμε όλα τα στοιχεία ώστε στο τέλος τέλος να μπορέσει να ε, αποτελέσει εποφελές έργο αυτό. Και θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε όσα απομένουν και στις τριμερείς αυτές διαπραγματεύσεις ε, να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλες αυτές τις πτυχές του κανονισμού. Ευχαριστώ. Οι σκιώδεις θέλουν να σχολιάσουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον εισηγητή για την, την εξαιρετική παρουσίαση του θέματος. Η ομάδα μου δεν έχει συγκεκριμένα πράγματα να θέσει ε, ως προς την συμφωνία αυτή. Οι διαπραγματεύσεις ε, ήταν θετικές. Πολλά από τα ζητήματα ωστόσο που έθεσε θα επανέλθουν ιδιαίτερα για το ζήτημα της πλατφόρμας. Στην ομάδα μου υπήρχαν επιφυλάξεις για, το, για την πρώτη της Επιτροπής να θεσπιστούν τέτοιες πλατφόρμες. Νομίζω ότι η μόνη καλή χρήση πώς το πω η χρηματοδότηση τέτοιων πλατφορμών δεν θα είναι εύκολη σε ό,τι αφορά τις, ε, προτεραιότητες, ε, τις προτεραιότητες αυτό θα είναι βασικό ζήτημα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο θα θέλει να διευκρινίσει και να εξειδικεύσει τις επενδυτικές προτεραιότητες στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στους κανονισμούς και τις διατάξεις ε, τους. Σε ό,τι αφορά ωστόσο το συγκεκριμένο περιεχόμενο δεν έχουμε, ε, τις δεν έχουμε προβλήματα, είμαστε ικανοποιημένοι. Κονέλη, Κορνέλη θες να προσθέσει κάτι? Ναι, σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Δεν είναι καθόλου απλό έργο να διαπραγματευτεί κανείς αυτά τα πράγματα όταν ταυτόχρονα χρονικά και τα θέματα του βασικού κανονισμού βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Συμφωνώ οπωσδήποτε ότι πάντα σε σύμφωνη γνώμη και συνενετικά πρέπει να προχωρούμε για να δούμε ποιες επιπτώσεις θα υπάρχουν σε σχέση με τον κανονισμό, από πλευράς κανονισμού για αυτά τα θέματα και πώς μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Και για τα θέματα της ε, ανάπτυξης των πόλεων ε, συμμερίζομαι αυτές τις θέσεις. Όμως ε, έχω επιφυλάξεις για την πλατφόρμα και είχα επιφυλάξεις από την αρχή. Το είπα επανειλημμένα, δεν με ικανοποιεί ιδιαίτερα η ιδέα μιας τέτοιας πλατφόρμας. Θα καλύτερα η Επιτροπή των Περιφερειών να είχε αναλάβει και να δημιουργούσε μια υποεπιτροπή. Δυσκολίες θα υπάρχουν και για τη χρηματοδότηση. Το ανέφερε ή αναφέρθηκε σχετικά ακροθυγός ο προλαλής σας και σε σχέση με τη, τη θέση τη, του εισηγητή ότι πρέπει να υπάρχει πρόσθετη αξία που θα απορρέει από αυτές τις δράσεις πρέπει νυφάλια να τα συζητήσουμε πραγματικά να υπάρξει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή την ε, κατεύθυνση ακόμα και εκείνοι που έχουν επιφυλάξει ε, σε σχέση με αυτήν πρέπει να γίνει λοιπόν καλή δουλειά προτεραιότητες για τις επενδύσεις ήταν σαφές ότι θα υπήρχαν προβλήματα και ότι θα είχαμε διακυμάνσεις Θέλω να πω συνολικά ότι τα σημεία τα οποία ήταν για μα σημαντικά για αυτή τη συζήτηση που κάποιε νέες πτυχέ, πολιτισμό, ε, δημιουργική οικονομία, πολιτισμό, culture, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα διατηρήσουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε αμάχη, να παραμείνουμε αμετακίνητοι διεκδικώντας τα. Τώρα, για τα, αυτά τα οποία είπε ο εισηγητή, σίγουρα σε αυτό το θέμα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι διαβουλεύσεις. Εξαρτάται και από την ικανότητα που θα έχουμε, διαπραγματευτική ικανότητα και φυσικά τα ιστορικού, ιστορικού χαρακτήρα κτίρια ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο. Δεν σταματά κάπου η αποδοτικότητα σε σχέση με την χρήση των ενεργειακών πόρων και θα υπήρχαν αρνητικές επιπτώσεις αν δεν υπήρχε βέλτιστη χρήση της ε, απόδοσης ε, αποδοτικότητας ενέργειας για αυτά τα κτίρια. Αν δεν μας πλήξει ε, ο χιονιάς και δεν έχουμε χιονοπτώσεις θα έχουμε καλές, καλή ευκαιρία να ξαναβρεθούμε και να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που καταβάλα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο για να θέσει κάποια ερώτηση. Ο κύριος Μετά την χθεσινή συζήτηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για τον καονισμό κοινών διατάξεων, είναι σαφές ότι η συζήτηση που γίνεται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί πραγματικά να ακολουθήσει αμέσως μετά τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Ο Γιάννη μας ότι έχουμε κάποιους θεματικούς στόχους. Είναι σαφές πάντως στη συζήτηση που βρισκόμαστε. Θέλουμε να εστιαστούμε στην αστική κινητικότητα από τη δική μας νοπτική γωνία, να μην αφαιρόμαστε ακριβώς υποδομές στο στόχο 4, αλλά μια νέα προσέγγιση. Η κινητικότητα είναι ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά επηρεάζει πάρα πολύ τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Συνδέεται άμεσα με την ρήπανση στις πόλεις. Επομένως θα πρέπει πραγματικά να επιμείνουμε στο ζήτημα αυτό και να μην δεχθούμε απλώς να γίνονται προτάσεις υποδομών οι οποίες μπαίνουν στο στόχο 4 στη συνέχεια. Πρέπει να εκφράσουμε κάποιες σαφείς ιδέες και πρέπει να δούμε ακριβώς τι θέλουμε στον στόχο υπαριθμών 7. Στη συζήτηση που είχαμε είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δεχόταν τις δικές μας τις απόψεις, αλλά άκουσαν πραγματικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε. Εμείς ε, δεν θέλουμε να μεταφέρουμε όλες τις βαριές υποδομές στον στόχο 4. Μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε να επιμείνουμε σε νέες ιδέες όπως η ευφύης πόλης ε, και το καθεξής και θέλουμε κατά αυτόν τον τρόπο να οργανώσουμε και τις ευφυείς αστικές μεταφορές. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να εμείνουμε σε αυτή μας τη θέση και ενδεχομένως να πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να αποσαφηνίσουμε την στάση μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως το ζήτημα αυτό. Έπειτα, το ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο Γιάνν. Στις πόλεις χρειάζεται ένα μείγμα μέσων, εργαλείων και πρέπει να γνωρίζουν έπειτα τα κράτη-μέλη πώς θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα αυτά. Χρειάζονται μια ευελιξία, μια ελευθερία στη χρησιμοποίηση των μέσων αυτών, γιατί καταλαβαίνετε ότι δίστανται πάρα πολύ οι καταστάσεις από τη μία χώρα στην άλλη. Άλλες χώρες ε, λειτουργούν με ένα σύστημα αποκέντρωσης, άλλες πάλι όχι. Επομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις ε, χρειάζονται απλώς κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, για άλλες χώρες θα χρειαζόταν όμως ένα ισχυρό νομοθετικό κείμενο. Όσον αφορά τώρα την αστική πλατφόρμα, Χθε θυμάστε ότι μιλήσαμε για την ε, ευφυή εξειδίκευση. Είχαμε μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό. Εξετάσαμε έπειτα το ζήτημα των περιφερειών εκείνων που θέλουν να επενδύσουν περισσότερο στην ευφυή εξειδίκευση, εκ των προτέρων μάλιστα, στα πλαίσια της αρχής της ε, αιρεσιμότητας. Και είδατε ότι 140 περιφέρειες ήδη έχουν καταχωρηθεί σε αυτό το κοινό κέντρο ερευνών της Σεβίλης και ουσιαστικά ηγούνται τις διαδικασίες αυτής. Έχουμε πάρα πολλές όμως προτάσεις. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε την πλατφόρμα αυτή. Πρόκειται απλώς για ένα λειτουργικό σχήμα το οποίο ευνοεί τη συνεργασία. Ας μην δημιουργούμε όμως νέες δομές οι οποίες τελικά σπαταλούν περισσότερα χρήματα. Στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής βλέπετε πραγματικά τι σημαίνει αστική επένδυση. Υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις που ήδη έχουν την εμπειρογνωμοσύνη ήδη βρίσκονται στην ηγεσία, στην πρώτη γραμμή πάρα πολλών προγραμμάτων. Από μόνες τους λοιπόν μπορούν να ολοκληρώσουν, να διεκπαιρεώσουν όλα αυτά τα προγράμματα. Ας μην δημιουργούμε λοιπόν νέες πλατφόρμες, ας μην δημιουργούμε νέες δομές. Ας αρκεστούμε στην υφιστάμενη συνεργασία η οποία έχει μια πολύ θετική δυναμική αυτή τη στιγμή. Γιάν, κινείσαι πάντως σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση, είσαι πολύ αποτελεσματικός στις, στους τριμερείς διαλόγους εκπροσωπείς πάρα πολύ καλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την εντολή που σου έχει δοθεί και θεωρώ ότι θα καταφέρουμε στα πλαίσια του κανονισμού γενικών διατάξεων να επιλύσουμε μέσα στους επόμενους μήνες τα εκκρεμή αυτά ζητήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει. Εφόσον λοιπόν καταφέρουμε να λύσουμε τα ζητήματα αυτά θα καταλήξουμε και σε μια κοινή συμφωνία. Αυτά είχα να σας πω. Συγχαρητήρια Γιάννα. Thank you. I if there are any άλλα σχόλια από τους βουλευτές, αλλά προς την Επιτροπή να στραφώ. Πρώτη ερώτηση, μας ακούτε? Μα και βέβαια σας, ακούμε, πάντα σας ακούμε. Ο τρίλογος ήταν πολύ χρήσιμο πλαίσιο για να διευκρινίσουμε μια σειρά θεμάτων και κάποιες παρα, παρεξηγήσεις και ορίσαμε και καλύτερα, ορίσαμε καλύτερα κάποιες από τις θέσεις Να αναφερθώ στα τέσσερα σημεία εντάχει. Πρώτον, το θέμα της εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε πόλεις. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο της πρότασης της Επιτροπής. Αυτό που ήταν χρήσιμο στον περίλογο αυτό ήταν ότι μπορέσαμε να προσαρμόσουμε το κείμενο στην πραγματικότητα, ιδίως δε να προβλέψουμε μεγαλύτερη ευελιξία στα επιχειρησιακά προγράμματα και στους παραδοσιακούς μηχανισμούς εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Το θέμα βέβαια της εκχώρησης αρμοδιοτήτων παραμένει ανοιχτό. Θα πρέπει να το συζητήσουμε στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Να πω και κάτι για την πλατφόρμα. Ήταν χρήσιμη συζήτηση στο Συμβούλιο. Διευκρινίσαμε το ρόλο της πλατφόρμας. Ο στόχος της δεν είναι να επικαλύψει τις δραστηριότητες υφιστάμενων μηχανισμών, δομών, οργανισμών. Έχουμε δύο νέα πράγματα στον οργανισμό. Πρώτον, μία εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε πόλεις όπως είπε ο εισηγητής, είναι ε, πιλωτικό αλλά περιλαμβάνει μεγαλύτερη εμπλοκή των πόλεων στα έργα αυτά και η προσέγγιση, ο στόχος αυτής της καινοτόμου προσέγγισης είναι για να μάθουμε. Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό που δεν χρειάζεται να είναι μεγάλος μηχανισμός αλλά θα επιτρέπει τη δικτύωση και θα, την τον καθοδηγεί επιτροπή όχι γιατί θέλουμε πάντα να το κάνουμε αυτό, αλλά γιατί νομίζουμε ότι η Επιτροπή είναι στην καλύτερη θέση να διδάσκεται από τα μαθήματα της διαδικασίας εκχώρησης ε, σε αρμοδιότητα και να διαδώσει τα θετικά τις δραστηριότητες αυτές. Στη συζητήση των λόγο επαναλαμβάνω προχωρήσαμε και καλύψαμε αρκετές από τις ανησυχίες που τέθηκαν στην Επιτροπή. Να πω δύο λόγια για τις δημιουργικές ε, βιομηχανίες, το, το, δημιουργικό κλάδο των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το μόνο που πρέπει να προσέχουμε είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε με τον κανονισμό. Ο κανονισμός, όπως ακούσατε κι εσείς, ε, είπατε κι εσείς, είναι ένα σημαντικό κείμενο για όσους προετοιμάζουν προγράμματα. Τώρα, αυτό το θέμα της έξυπνης εξειδίκευσης. Στο κέντρο της νέας προσέγγισης προς την καινοτομία, την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την έρευνα, πρέπει να υπάρχει κάτι που συνδέεται με τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιφερειών. Οι επιλογές που γίνονται σε κάθε περιφέρεια θα γίνονται βάσει της ανάλυσης που κάνουν οι ίδιες. Η έξυπνη εξειδίκευση προτάθηκε γιατί από τα προηγούμενα διδάγματα ε, διαπιστώσαμε ότι οι δημιουργικέ βιομηχανίε είναι καλέ για όλου. Η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία ε, είναι θετική για όλου. Και πιστεύουμε ότι αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε με αποτελεσματικό τρόπο αν έρχονται από σωστή ανάλυση τη κατάσταση από τι ίδιε περιφέρειε. Γι' αυτό είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί ε, στο να εισάγουμε στον κορονομισμό συγκεκριμένου κλάδου, Όχι διότι δεν πιστεύουμε ότι πολιτιστική βιομηχανία σε πολλές περιοχές δεν θα συμβάλλει στην αύξηση της ανάπτυξης. Όχι. Πιστεύουμε ότι τούτο πρέπει να είναι ε, συνέπεια της διαδικασίας συζητήσεων στην Επιτροπή εκ των κάτω προς τα άνω. Μία τελευταία παρατήρηση για την ε, μεταφορά της βιώσιμης αστικής τεχνολογίας. Εδώ ακριβώς μπορέσαμε να μπούμε σε λεπτομερέστερη συζήτηση όταν συζητούσαμε τον κανονισμό του Ταμείου, του Περιφερειακού Ταμείου και εδώ νομίζω είναι αρκετά σαφή η θέση των τριών θεσμικών οργάνων. Για να απαντήσω στην Πρόεδρο, η τρίλογη ήταν χρήσιμο πλαίσιο για να μπορέσουν οι τρεις ε, θεσμοί να μ' ακούσουν και να καταλάβουν ένα τον άλλον. Για αν θέλεις να ολοκληρώσει τη συζήτηση? Ναι. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Δεν υπάρχουν μεγάλες διχογνωμίες όπως βλέπετε. Ορισμένα από αυτά που αναφέρθηκαν ωστόσο θέλω να τα σχολιάσω. Πρώτον, η πλατφόρμα Urban, η αστική πλατφόρμα, η εντολή και η θέση μας ήταν ε, από πλευρά Κοινοβουλίου αρνητική. Δεν χρειαζόμασταν, λέμε, νέες αρχές, ε, νέα Airbact που στην ουσία επικαλύπτει και ξανακάνει αυτά που έκανε η Airbact. Δεν χρειαζόμαστε Αυτό που δυστυχώς εκφράστηκε από τους εκπρόσωπους της Επιτροπής, χρειαζόμαστε ένα πολιτικό όργανο η Επιτροπή, γι' αυτό δημιουργήθηκαν πολλές παρανοήσεις. Μετά τις διευκρινήσεις ωστόσο από την Επιτροπή ότι αυτή η δράση έχει σε στόχο να επαληθεύσει κατά πόσον η δράση αυτή δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τα ουσιαστικά κονδύλια από την τεχνική βοήθεια που θα εξετάσει αν λειτουργεί όχι ιδίω ε, για το 5% της καινοτόμης δραστηριότητας και μόνο από αυτό χωρίς να υπάρχει νέο όργανο που θα δημιουργείται ΣΑΗ αλλά μόνο ως τεχνική βοήθεια και ανταλλαγή εμπειριών. Νομίζω ότι αυτό πλέον είναι σαφές. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες επενδύσεις, εμείς βεβαίως θα υποστηρίξουμε τις θέσεις μας. Είναι γεγονός ότι όταν βλέπετε τις επενδυτικές προτεραιότητες και όταν θέλουμε να τις κάνουμε γενικές χωρίς να αναφέρουμε κανέναν κλάδο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς όμως τις προτεραιότητες αναφέρουμε κάποιους κλάδους. Και όσο Κάποια αναφέρουμε, κάποια δεν τα αναφέρουμε. Αυτά που δεν αναφέρουμε δεν υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Γι' αυτό ορισμένα από τα στοιχεία θα ήταν σκόπιμο να τα βάλουμε στο κείμενο. ακόμα και κάποια πράγματα που μπορεί να μην τα δεχθεί καθόλου το Συμβούλιο. Πιστεύω ότι ορισμένα σημεία πρέπει να αναφέρουμε ρητά και να τα υποστηρίξουμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Τούτο ωστόσο δεν αλλάζει τη γενική στάση, η ατμόσφαιρα στον τρίλογο ήταν πολύ καλή και θετική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν χρειάζεται να πάρουμε απόφαση. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 12 της μερίσιας διάταξης, έκθεση του Βίκτορ Μποστινάρου για το Ταμείο Συνοχής. Σε ευχαριστώ, Ντανούτα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχω σπουδαία πράγματα να σας πω αυτή τη στιγμή, γιατί είχαμε μόνο έναν τριμερή διάλογο, όπως το γνωρίζετε. Και κατά τη διάρκεια του τριμερούς αυτού του διαλόγου τα πράγματα εξελίχθηκαν καλά. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια βασικά σημεία, τα οποία συζητήθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση και για τα οποία είχε επιτευχθεί συμφωνία. Άρθρο υπαριθμών 2. Ένα από τα βασικά σημεία είναι το ακόλουθο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε υποβάλει μια τροπολογία για να συμπεριληφθεί στο άρθρο 2 και μια αναφορά στην διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, εφόσον κάποια χρήματα θα μεταφερθούν από το Ταμείο Συνοχή στο ε, CF η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για διαφορετικούς λόγου έκαναν τις ακόλουθες προτάσεις. Το Συμβούλιο μας είπε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία επ' αυτού και δεν έχουν εντολή για να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε όμως εμείς είναι ότι στο Συμβούλιο υπάρχει ακόμα μία αντίθεση στο CEF, στη διευκόλυνση δηλαδή συνδέοντας την Ευρώπη, και αυτό δημιουργεί ανησυχίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει μετάθεση αυτή κονδυλίων. Έτσι λοιπόν, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουμε ότι έχουμε την απαραίτητη ευελιξία και ότι προσπαθούμε τελικά να βρούμε μια συμβαστική λύση η οποία θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε τα κονδύλια αυτά στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής προκειμένου να καλύπτονται συγκεκριμένες περιφέρειες και κράτη-μέλη. Έκκλησή μου προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι αν τελικά αποδεχθεί η Επιτροπή τη μεταφορά των κονδυλίων αυτών, τότε προφανώς θα πρέπει να γίνει μια αναλλαγή όσον αφορά το CF στον κανονισμό του Ταμείου Συνοχή, Αυτή είναι η εντολή που έχουμε εμεί, Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δεχθεί πάντω τη μεταφορά αυτή. Κι αν ο ίδιος κανόνας τελικά υπάρξει και στον κανονισμό γενικών διατάξεων, αλλά και στον κανονισμό της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη, τότε πραγματικά αυτό θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως το σημαντικότερο νομικό επιχείρημα για να πούμε ότι το CF θα πρέπει τελικά να υλοποιηθεί, να γίνει πραγματικότητα. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξο και πιστεύω ότι με την Ιρλανδική Προεδρία θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμβαστική λύση. Πρέπει πάντω εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πούμε ότι έχουμε προχωρήσει περισσότερο, είμαστε πιο ευέλικτοι και είμαστε σε θέση τελικά να προτείνουμε μια ρεαλιστική λύση για κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Όσον αφορά κάποιες διατάξεις που εξαιρούν κάποιες δραστηριότητε που καλύπτονται από το ETS, εδώ πέρα η στάση μα είναι ίδια με το Συμβούλιο. Η συμπαραγωγή θα πρέπει να είναι επιλέξιμη με την εξαίρεση εκείνων των μονάδων παραγωγής που ξεπερνάνε τα 20 ΜΒ. Συμφωνία από αυτού υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και αυτό είναι θετικό. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα κάποια προβλήματα, τα οποία θα εξετάσουμε και αργότερα, όταν θα μιλήσουμε για τις επενδυτικές προτεραιότητες που έχει υποβάλει στο άρθρο 3 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, η δυνατότητα ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς επίσης και την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια, την ίδια τροπολογία έχουμε εδώ πέρα με το Συμβούλιο, επομένως έχει διατηρηθεί. Για το άρθρο 3. Επενδυτικέ προτεραιότητε. Τα βασικά σημεία είναι τα ακόλουθα. Το Συμβούλιο θα υποβάλει μια πρόταση προκειμένου να συμπεριληφθεί με άλλη διατύπωση αλλά με το ίδιο νόημα το ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα πρέπει αυτέ κατά προτεραιότητα να αποφεληθούν από την στήριξη για την ενεργειακή αποδοτικότητα και για την χρήση ανανόσιμων πηγών ενέργεια. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι οι μόνες. Νομίζω ότι η λύση αυτή είναι αρκετά ευέλικτη και τελικά καλύπτει και τις δύο πτυχές, και τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις ανάγκες όλων των άλλων. Τώρα, η επενδυτική προτεραιότητα για την ανανεώσιμη χρήση ενέργειας στα κτίρια βρίσκει σύμφωνο και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει υποβληθεί η ίδια τροπολογία. Όσον αφορά τώρα το τομέα του ύδατος, το Συμβούλιο θεωρεί εδώ πέρα ότι η δική μας πρόταση είναι κάπως περιοριστική. Επίσης, Μέσω μια νέα διατύπωση πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε τόσο στι ανησυχίε του Συμβουλίου όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να πιστεύω πάντω ότι και οι δύο πλευρέ, και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μα βοηθήσουν να βρούμε τελικά μια συμβαστική λύση. Το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε έχει να κάνει με το ότι και η Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι κατά τις τραπολογίες μας που έχει να κάνει με την επενδυτική προτεραιότητα για την συμπαραγωγή καθώς επίσης και την υψηλή διανομή ενεργειακής ε, ε, αποτελεσματικής θέρμανσης. Το Συμβούλιο είναι κατά τη πρόταση αυτή γιατί θεωρεί ότι αν δημιουργηθεί επενδυτική προτεραιότητα για το ζήτημα αυτό, τότε θα αποκλειστούν άλλε επενδυτικέ προτεραιότητε που δεν αναφέρονται. Αποφασίσαμε να επαναφέρουμε το ζήτημα αυτό στην πραγματευτική ομάδα προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση. Έκτοτε, μέσω άτυπων συναντήσεων που είχαμε όλους σκιώδεις ε, εισηγητές, είπαμε όλοι μας ότι θα πρέπει πραγματικά να υποστηρίξουμε εκ νέου την εντολή που μας δόθηκε το καλοκαίρι. Ελπίζω λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμερούς διαλόγου θα καταφέρουμε να τονίσουμε τη σημασία του ζητήματος αυτού, γιατί είναι σαφές για όλα τα κράτη-μέλη της συνοχής ότι όταν θέτουμε τον στόχο της ε, υψηλής αποδοτικότητας της θέρμανσης και της συμπαραγωγής, τότε πραγματικά βοηθάμε και τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη και τις κοινότητες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές. Τους βοηθάμε όμως κιόλας να εξοικονομήσουν ενέργεια, να βελτιώσουν το μείγμα ενέργειας το οποίο χρησιμοποιούν και να φτάσουν τελικά σε ένα στόχο βιώσιμης ανάπτυξης ως προς την ενέργεια. Νομίζω λοιπόν ότι η συνεισφορά μας αυτή μέσω του στόχου αυτού θα συμβάλλει πάρα πολύ και στην αστική ανάπτυξη την οποία συζητούσαμε. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι στις 18 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που γίνανε στο Συμβούλιο για το ζήτημα αυτό, ορισμένα κράτη-μέλη είπανε σαφώς ότι είναι υπέρ της πρότασης αυτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω λοιπόν ότι το μήνυμα αυτό θα ακουστεί ξεκάθαρα και στεναρά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το σύνολο του Συμβουλίου. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ήμουν κάπως απογοητευμένος όταν είδα ότι το Συμβούλιο αντιτίθεται στο ζήτημα αυτό, στη δική μας την πρόταση, χωρίς όμως να έχει κάνει κάποια συζήτηση πριν. Αυτό πραγματικά με στενοχώρησε. Ένα άλλο τώρα σημαντικό σημείο που βασικά είναι και το ουσιαστικό μας συμπέρασμα. Αποφασίσαμε μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες οι διατάξεις και όλοι οι κανονισμοί που έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας για τις κατοικίες καθώς επίσης και όλες οι διατάξεις που έχουν να κάνουν με την αποδοτική θέρμανση που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής να έχουν τελικά την ίδια σειρά, την ίδια παρουσίαση προκειμένου να μην υπάρχει καμία σύγχυση, να έχουμε ακριβώς τις ίδιες διατάξεις για τα ζητήματα αυτά και στα δύο ταμεία. Μία τελευταία τώρα παρατήρηση, η οποία συνδέεται με το γεγονός ότι ο επόμενος τριμερής διάλογος θα εστιαστεί σε αυτό. Οι περίφημοι κοινοί δείκτες, στους οποίους αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Γιάννα είναι σημαντικό να αποφασίσουμε για το ζήτημα αυτό πολύ νωρίς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ο αντίκτυπος θα είναι σημαντικός και για το Ταμείο Συνοχής και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως είπαμε, δύο είναι εναλλακτικέ εκτελεστικές πράξεις και πράξεις εξουσιοδότηση. Και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να λέει ότι χρειάζεται πιο ελαστικές εφαρμοστικές πράξεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τουλάχιστον να μπορέσει να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ποια λύση είναι καλύτερη Εφαρμοστικές πράξει ή κατεξοδότηση πράξη. Αν προχωρήσουμε γρήγορα στο ζήτημα αυτό, θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια συμφωνία και με το Συμβούλιο. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει διχογνωμία αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο υπάρχουν κρατημέλη τα οποία αντιτίθενται στις κατεξοδότηση πράξεις. Θεωρούν ότι είναι πολλές. Τώρα, τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο επόμενος τριμερής διάλογος προβλέπεται για τις 27 Φεβρουαρίου. Εμείς είχαμε προτείνει να γίνει ένας ε, τριμερής διάλογος στην επόμενη Ολομέλεια του Στρασβούργου, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά μας αυτό εξαιτία των ε, υποχρεώσεων που έχει τόσο το Συμβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντω, ξεκολουθώ και πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου έχοντα κατά νου και την πραγματικότητα ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν πραγματικά προβληματικά σημεία, δεν υπάρχει διχόνοια για ουσιαστικά σημεία, πιστεύω ότι μέχρι, το, μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα έχουμε ολοκληρώσει τον κανονισμό του Ταμείου Συνοχή, θα είναι έτοιμο το κείμενο και ουσιαστικά θα περιμένουμε να εγκριθούν όλα αυτά τα σημεία που περιέχει ο κανονισμό. Ευχαριστούμε πολύ, Βίκτο. Κορνέλια, θα ήθελε να σχολιάσει η μόνη σκιώδη που παρίσταται. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Είναι σαφές υποστηρίζουμε τον εισηγητή στο θέμα της διασύνδεσης της Ευρώπης, Connecting Europe. Πρέπει να παραμείνουμε σκληροί σε αυτό το θέμα. Με σκληρή μάχη πετύχαμε αυτή τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου και δεν μπορούμε να την απεμπολίσουμε, να την εγκαταλείψουμε. Εντάξει για συμβιβασμού, έστω, αλλά πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην θεμελιώδη αυτή πτυχή του θέματος, να μείνουμε πιστοί. Δεύτερη παρατήρηση για το συνολικό θέμα ενεργειακής αποδοτικότητας και το συνολικό θέμα των της ενέργειας. Να προσέξουμε ιδιαίτερα εδώ, να μην έχουμε διαφορετικές τοποθετήσεις για αυτό το θέμα στα διαφορετικά ταμεία. Δεν μπορεί κανείς να οπισθοχωρήσει και να δεχθεί κάτι λιγότερο. Πρέπει να υπάρξει σαφής ένταξη των ταμείων σε αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω από τη θέση που υιοθετήσαμε και εκπονήσαμε. Είναι αποφασιστική σημασία οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να μπορέσουν να προαχθούν. Η συμπαρα... συμπαραγωγή να το ξανασυζητήσουμε εντάξει, να δούμε, να καταλήξουμε σε μια θετική έκβαση αν είναι δυνατόν. Και ένα άλλο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατά πόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Πάντα λέγαμε ιδιαίτερη προσοχή να στρέφουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό λοιπόν δεν επιτρέπεται να υπαναχωρήσουμε σε αυτό ή να το αμελήσουμε. Κατά τα άλλα συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε ε, Φανίστερ Ρόι. Σύντομα ε, συγχαρητήρια για αυτή την πρόοδο. Η προσωπική μου αντίδραση ποια είναι. Είναι να πω ότι σε σχέση με το Ταμείο Συνοχής και αυτούς τους στόχους που έχει προσπαθεί να εντάξει το Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με τη συμπαραγωγή και τον τομέα της στέγασης, πραγματικά δίνουμε τεράστια προώθηση σε αυτά που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως στόχους της στρατηγικής για το 2020 και για το, τη συνοχή συνολικά και τις διαβουλεύσεις και συζητήσεις. Η παρατήρηση ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ελαστικότητα, αλλά να δούμε τι θα γίνει εδώ για αυτό το χαρτοφυλάκιο τελικά του κυρίου Έτιγκερ. Και στο χαρτοφυλάκιο της κυρίας Χέντεγκαντ για το περιβάλλον. Εκεί που πρέπει να εστιαστούμε είναι μεγαλύτερη επικοινωνία. Να διαπραγματευτούμε, αλλά να έχουμε και καλύτερη επικοινωνία, ώστε να γνωρίζουν, ώστε να γνωρίζουν ότι το Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής περισσότερο προς αυτή την επίτευξη αυτής της αρχιτεκτονικής για τους στόχους του 2020, με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτό κάνει το Κοινοβούλιο, με άλλα λόγια αναζητούμε καμιά φορά αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα να υπάρξει αλλού κάποιο περιθώριο ελιγμών ε, μέσω άλλων κονδυλίων ή άλλων δράσεων. Αυτό δείχνει όμως τη δέσμευσή μας, έτσι, να προχωρήσουμε. Και επειδή οι τριμερείς διάλογοι εξελίσσονται βήμα προς βήμα, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να επικοινωνούμε επ' αυτού του θέματος, να περνάνε τα μηνύματα του Ευρωκοινοβουλίου αποτελεσματικά. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Προτού δώσω τον λόγο στον Πίτερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να ζητήσω Πίτερ, θα μπορούσε στα επιχειρήματα αυτά τα οποία ε, είχαν παρουσιαστεί, νομίζω ήταν σε σχέση με το γενικό κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, στο τριμερή διάλογο, σε σχέση με το κεκτημένο για το νερό για το πόσιμο νερό γιατί έχουμε το πρόβλημα ότι προστίθενται εδώ περισσότερα στοιχεία και η θέση της Επιτροπής είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ε, η ε, δυναμική του κεκτημένου και ότι θα πρέπει αυτές οι πτυχές να μπορούν έτσι να αντιμετωπιστούν. Μπορείς να πεις δύο λόγια γι' αυτό. Ευχαριστώ. Πρώτα εντάχει να πω ότι συμμερίζομαι την αξιολόγηση, την εκτίμηση του εισηγητή όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους, όσον αφορά την διατύπωση, το κείμενο και για τον τομέα του νερού και για τον τομέα των αποβλήτων. Η, το μέλημα, η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι ίσως η πρόθεση του Ευρωκοινοβουλίου δεν αντανακλάται υποχρεωτικά υπαρκώς στα κείμενα. Και στις δύο αυτές λοιπόν περιπτώσεις, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία για τα απόβλητα και η οδηγία πλαίσιο για το νερό, και σε σχέση με τα, τη διαχείριση ε, ποτάμιων, λεκανών ουσιαστικά αφορούν όλες τις επενδύσεις και δράσεις για αυτούς τους τομείς. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πρόβλημα αν ένα κράτος μέλος ήδη σήμερα υλοποιεί όλες αυτές τις διατάξεις και προδιαγραφές και θέλει να πάει ακόμα πιο πέρα. Θα ανησυχούσε όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δημιουργούσαμε μια παράλληλη πορεία παράλληλη διαδρομή για θέματα τα οποία δεν αποτελούν τμήμα του νομοθετικού πλαισίου όσοι υφίσταται σήμερα. Η ιδέα να υπάρξουν επενδύσεις για τον τομέα του νερού που δεν θα βρίσκονται στο πλαίσιο της, ε, των ε, προγραμμάτων διαχείρισης των ποτάμιων λεκανών είναι κάτι που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να δεχθούμε. Ανοίγει η δυνατότητα εδώ να υπάρχουν ασύμβατα πράγματα σε σχέση με το κεκτημένο. Η ιδέα μας είναι ότι με κάποιες αναδιατυπώσεις ε, μπορούν αυτά να αποσαφινιστούν, να διευκρινιστούν, ότι το βασικό κείμενο είναι το νομοθετικό σχετικό κείμενο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν έχουμε πέρα από τις βασικές ε, τέτοιες ε, απαιτήσει κάτι από τα κράτη-μέλη τότε θα μπορεί να γίνεται αυτό, θα επιτρέπεται. Κάποιες ε, δύο παρατηρήσεις ε, για το θέμα της ε, διευκόλυνσης του μέσου για τη διασύνδεση της Ευρώπης. Υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι θέμα μόνο διατύπωσης του κειμένου. Δεν είναι θέμα ουσίας περιεχομένου. Είναι σαφές για αυτή τη συμφωνία, κατανοούμε τους στόχους και τη συμφωνία όπως θέλουμε να λειτουργήσει. Θα έχει επιπτώσεις όσον αφορά τους κανονισμούς του Ταμείου. Μια και πρόκειται για το CPR, εκεί θα πρέπει να στοχεύει. Δεν είναι θέμα όμως επίμαχο αυτό, είναι θέμα διατύπωσης ακριβώς και ορολογίας. Όπως είπα επανειλημμένα στο παρελθόν, έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις να ανοίξει το Ταμείο Συνοχής για την, αποδοτικότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα στη στέγαση. Νομίζουμε ότι εδώ ε, θα ήταν κάτι το οποίο υπό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα μπορούσε να ενταχθεί. Όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άλλες απόψεις και μάλιστα ισχυρές ε, ε, θέσεις, απόψεις με επιχειρήματα από άλλους γι' αυτό. Τώρα για τη συμπαραγωγή και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με άλλα λόγια και θέρμανσης υπό τις προτεραιότητες προτεραιότητε για τι επενδύσει, Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εξεύρουμε μια λύση για αυτό το θέμα μέσα στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων. Σας ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ. Βίκτορ, άλλα σχόλια. Χαρούμενος ε, φαίνεσαι, αλλά θέλεις να σχολιάσεις πάντως. Όχι να σχολιάσω. Με ενθαρρύνει η δήλωση του κ. Πέτκοβιτς και πραγματικά νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να τον ευχαριστήσω προσωπικά και τη Γενική Διεύθυνση περιφερειακή Αναπτύξη για τον επικοδομητικό τρόπο τον οποίο δουλεύουν για την επίτευξη της αναγκαία συμφωνίας όταν χρειάζεται. Τα συμπεράσματά μου είναι τα ίδια. Δεν υπάρχει συμφωνία για τίποτα όσο δεν υπάρχει συμφωνία για όλα. Η ανάγκη συμβιβασμού πρέπει να εκφράζεται και να επιβεβαιώνεται από κάθε έναν από τους τρεις εμπλεκόμενους. Και λαμβάνοντα υπόψη τα στρατηγικά θέματα. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν τα ίδια συμφέροντα, δεν έχουν, μπορεί να έχουν και το ίδιο όραμα. Πιστεύω θα το πετύχουμε. Με την ίδια ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις. Πραγματικά με εντυπωσίασε η εξαιρετικά θετική ατμόσφαιρα συνεργασίας που είχαμε και η κοινή μας προσέγγιση, για να μην πω το κοινό μας όραμα, για το πώς θα έπρεπε οι περιφέρειες ε, και τα κράτη-μέλη της συνοχής να ξοδεύουν, να δαπανούν τις δαπάνες της συνοχής. Με το τελευταίο σχόλιο του Πίτερ είμαι ακόμα πιο προσεκτικά αισιόδοξο και ευχαριστώ τον Λαμπέρτ για την ιδέα να προωθήσουμε αυτό που κάνουμε εδώ για κάτι που είναι ουσιαστικό για τη στρατηγική ενόψη του 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Βίκτορ. Βάστα μικρό καλάθι λέμε. Εμείς λέμε ότι μας ικανοποιεί αυτό που κάνει η Βιτοπή για να τη σπρώξουμε να κάνει κι άλλα. Κλείνω νομίζω. Και πάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία, οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν καλά κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Αν θέλουμε τώρα να υπάρξει πρόοδος στην Άνοιξη, γρήγορη πρόοδος, ιδίως για το γενικό κανονισμό, βλέπουμε ότι οι προθεσμίες πιέζουν. Εάν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι το Μάρτιο-Απρίλιο, θα πρέπει να συμφωνήσουμε περισσότερες ε, συνεδριάσεις στους επόμενους μήνες. Έχουμε μία συνάντηση το Φεβρουάριο αλλά η διαπραγματευτική ομάδα στο Κοινοβούλιο είναι πρόθυμη να προχωρήσει περαιτέρω και ταχύτερα για τα τεχνικά θέματα. Τι μπορούμε να πούμε. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα όπου θα εξετάσουμε τα θέματα 5, 6, 7, 5, 6, 17, 18 και 19. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνία για τα άρθρα αυτά και τα γρήγορα ούτως ώστε να μιλήσουμε για το περιεχόμενο του άρθρου αυτού, των άρθρων αυτών γρήγορα. Θα το δούμε λοιπόν τη Δευτέρα με την ομάδα για να ξεκινήσουμε συζητήσεις ε, ως προς το περιεχόμενο. Πριν τα Χριστούγεννα επί Κυπριακής Προεδρίας μπορέσαμε να ασχοληθούμε με το άρθρο 2, με το άρθρο 2 τους σκοπούς της περιφερειακής συνεργασίας, το 7 για το περιεχόμενο των προγραμμάτων, το άρθρο 8 για τις κοινέ δράσεις, το άρθρο 11 για την επιλογή των δράσεων και το 12 για τους δικαιούχους. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα άρθρα μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχε πραγματική διαφωνία στο Συμβούλιο. Μπορούσαμε να έχουμε θετική συμφωνία και να τηρήσουμε την εντολή που λάβαμε από την Επιτροπή. Ωστόσο, περιμένουμε το έγγραφο των τεσσάρων στυλών για να δούμε όλα τα θέματα ένα προς ένα. Ελπίζουμε ότι τούτο θα είναι σύμφωνο με, τις γενικές, με τη γενική εντύπωση που είχαμε μετά τις διαπραγματεύσεις. Είδαμε, είδε το Συμβούλιο τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, είδαμε τα θέματα των υποδομών, την ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ εργαλείων, Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε καλή συμφωνία με το Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Εμείς ε, δεσμευόμαστε εν μέρη από τους κανονισμούς γενικής, του, από το γενικό κανονισμό και μπορέσαμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων βασίζονται στις ε, συμβιβαστικές προτάσεις που πετύχαμε για τα προηγούμενα άρθρα. Κοιτάμε να δούμε ποιες αποφάσεις θα ληφθούν για τα υπόλοιπα άρθρα. Οι δυνατότητες τώρα των τρίτων χωρών να λειτουργήσουν ως leaders σε συγκεκριμένα έργα. στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Ε, αυτό είναι πιο προβληματικό, αλλά νομίζω ότι και εδώ θα υπάρξει συμφωνία με το Συμβούλιο. Για συγκεκριμένα θέματα, στο άρθρο 2 υπήρχε μια μακρά συζήτηση για τον ορισμό της, ε, του interactive, του διενεργού. Το Συμβούλιο ήθελε να περιορίσει την εμβέλεια του ορισμού αυτού. Από ό,τι ωστόσο ακούω, το Συμβούλιο είναι έτοιμο να δεχθεί τον ορισμό της διαλειτουργικότητας όπως τον προτείνει το Κοινοβούλιο. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν ε, νομίζω προχωρούν καλά μέχρι τώρα. Θα υπογράμμιζα εκ νέου ότι δεν υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και θα εξετάσουμε ιδιαίτερα τα θέματα των επενδυτικών προτεραιοτήτων και θεματικά ζητήματα, με μακρά συζήτηση προφανώς που σχετίζεται, σχετίζεται πολύ με το CPR. Αυτά προς το παρόν. Ελπίζω ότι η αργότερη επιτροπή θα μπορέσει να, μπει, να μπούμε και σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ευχαριστώ. Μάρι Τερέζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις θέλω να ευχαριστήσω τη Ρίκα Μανέρα για την ατμόσφαιρα που κατάφερε να περάσει στην ομάδα οι διαπραγματεύσεις γίνονται εξαιρετικά θετικέ, ε, είναι, προχωρούν εξαιρετικά γρήγορα, με καλή ατμόσφαιρα. Πολλά μένουν εκκρεμή ακόμα, είναι αναμονή του τέλους των διαπραγματεύσεων. Ανάλογα βέβαια με το πώς προχωρά ο γενικός κανονισμός του Περιφερειακού Ταμείου, προχωρούμε και εμείς. Προφανώς η εδαφική συνεργασία πρέπει να συντονίζεται με τα υπόλοιπα ταμεία, είναι προφανές αυτό. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδίως ε, τον ε, ειδικό χαρακτήρα της περιφερειακής συνεργασίας. Προφανώς πρέπει επίσης να το απλοποιήσουμε και να το προσαρμόζουμε για να έχουμε και οικονομίες κλίμακας και για να μπορεί να είναι ανταγωνιστική η περιφερειακή δραστηριότητα. Ένα σημαντικό προφανώς στοιχείο είναι οι διαπραγματεύσεις του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σήμερα το πρωί είχαμε μια συνάντηση της ε, διασυνοριακής ομάδας επαφής θέλω να σας ε, ενημερώσω και προσοχή. Ε, υπάρχει κίνδυνος από τις περικοπές στην πολιτική συνοχής, ιδίως δε στην ε, περιφερειακή συνεργασία, να ε, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιβράδυνση στις δικές μας πολιτικές, ιδίως στην περιφερειακή, στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία. Πρέπει να προχωρήσουμε για να υπερασπιστούμε τον προπολογισμό που στην τελευταία πρόταση του Χέρμαν Βαν Προμπάι είχε περικοπεί κατά 25%. Και θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους, από όλα τα κράτη-μέλη, να ε, τονίσετε, να πιέσετε για την σημασία της πολιτικής αυτής. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και για την εικόνα ακόμα της Ένωσης στους πολίτες να αναπτύξουμε την πολιτική αυτή γιατί δίνει συγκεκριμένη, ε, συγκεκριμένη εικόνα για την Ευρώπη. Ε, σήμερα το πρωί ε, θα ακούσουμε τον κύριο Λαμασούν, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Προσοχή, αυτά που μας λέει είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Ευχαριστώ. Ο Φρανσουά Αλφόνση. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπε η Μαρή οι διαπραγματεύσεις προχωρούν όντως παρότι ε, τρενάρουν σε ορισμένες φάσεις, έτσι είναι η ζωή. Θα πρέπει προφανώς να αυξήσουμε τις συναντήσεις, τον αριθμό των συναντήσεων και μην ξεχνάτε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές εξαρτώνται από άλλα θέματα, τον γενικό κανονισμό και τις δημοσιονομικές προοπτικές, όπου πραγματικά η κατάσταση είναι ανησυχητική. Υπάρχει κάθε κυβέρνηση, κάθε κράτος στα πλαίσια της ε, διαδικασίας ομοφωνίας θέτει τις δικές της κόκκινες γραμμές. Δεν αγγίζεται αυτό, δεν αγγίζεται εκείνο, δεν αγγίζεται το άλλο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πετύχουμε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μετατρέψει την εδαφική συνεργασία σαν δική του κόκκινη γραμμή για τη διαπραγματεύσει. Γιατί αλλιώ έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ όμορφο κανονισμό, εξαιρετικού στόχου, χωρί λεφτά. Ο Γιάννη Νίλσον. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι αισιοδοξία από αυτή την επίστολη μπορώ να ερμηνεύσω και αυτό θα μπορούσε να έχει θετική έκβαση αν πράγματι ισχύει. Το ερώτημά μου αφορά την μακροπεριφερειακή στρατηγική. Είναι ενδιαφέρον. Αν δεν κατανόησα τα όσα αναφέρθηκαν Αναφέρεται ότι η διασύνδεση είναι σαφή στα περιφερειακά προγράμματα θα πρέπει να καλύπτονται με αυτόν τον τρόπο και να συνεισφέρουν για τη μακροστρατηγική, μακροπεριφερειακή στρατηγική, ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί και να χρηματοδοτείται. Ισχύει πράγματι αυτό. Διασύνδεση με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Ευχαριστώ. Ναι, Απλά ήθελα να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου στην παρατήρηση του συναδέλφου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ε, σήμερα το πρωί είχαμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που είπε ότι είναι ενδιαφέρον αν έχει κανείς λιγότερα ή περισσότερα κονδύλια για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Θα ήθελα να δραχθώ της ευκαιρία σε σχέση με αυτή τη συζήτηση. Καθότι γνωρίζω δεν υπάρχουν κονδύλια για την μακροπεριφερειακή προσέγγιση σύμφωνα με τη σουηδική πρόταση υπάρχει πιθανότητα, η δυνατότητα από το Interreg 2 να χρησιμοποιηθούν ε, στοιχεία για την ενίσχυση, υποστήριξη ενώ συζητούμε λοιπόν τα θέματα αυτά τα διαμεθοριακά ή θα συμπεριληφθεί η διαπεριφερειακή διαπεριφερικη συνιστοσα και θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα ή θα ακολουθήσουμε την ίδια πορεία. Θα είναι η πρόσθετη ε, αξία η συνεργασία, αλλά χωρίς κονδύλια για την υποστήριξη. Πρέπει να είναι σαφές αυτό, να αποσαφινιστεί σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την τοποθέτησή της, γιατί διαφορετικά αυτός ο κανονισμός ε, θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Πώς θα λειτουργήσει, αν κάποιος για τις μακροπεριφερειακές αυτές προσεγγίσεις σε σχέση με τα όσα ανέφερε η Μαρή Τερέζ πάρει κάτι δεν θα παραμείνει τίποτα για τη διασυνοριακή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λάμπερτ Φανίστερ Ρόι. Λάμπερτ Φανίστερ Ρόι, παρακαλώ. Thank you, thank you very much, Ευχαριστώ πολύ για το θέμα που, τη, της Ρίκα. Ρίκα παρακολουθείς παρακαλώ αυτά που λέω. Παρακολουθείς εντάξει. Για την παρατήρηση που έκανες για τον προϋπολογισμό θα έλεγα πραγματικά στην εντολή μας και με τα όσα συζητήσαμε χθε, όπως τα συζητήσαμε υπό, με την παρουσίαση της Ιρλανδικής Προεδρίας, αναφέρθηκε ότι ήθελαν να σεβαστούν πλήρως τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Και θα έλεγα για αυτό το τμήμα διατυπώσαμε εμείς πρόταση 5%. 5% των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Δεν θα έπρεπε να μετακινηθούμε καθόλου από αυτό το αίτημα, από αυτή τη διεκδίκηση. Άσχετα ποια θα είναι η έκβαση για τα μάκρο ε, θέματα προσέγγισης. Παραμένουμε στο 5%. Ως προτεραιότητα πρέπει να παραμείνουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα ως διεκδίκηση. Διότι τι θέλουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε με σωστό τρόπο αυτή την ε, πορεία. Διασυνοριακή συνεργασία. Εντάξει, πρέπει να ε, χρηματοδοτείται και πρέπει να διασφαλιστεί αυτό. Είναι η, εδαφική, η θέση για την εδαφική συνεργασία που μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Η Ευρώπη, όπως τη συζητήσαμε χθε για την ευφυή εξειδίκευση, smart specialization. Γοργά μπορεί να πετύχει πολλά θετικά αποτελέσματα με καλύτερη συνεργασία η Ευρώπη. Είχαμε προγράμματα για τη διάχυση γνώσης, ε, πάσης φύσεως προγράμματα και δράσεις και αυτά έχουν πολύ περισσότερες επιπτώσεις, ευρύτερες επιπτώσεις από ό,τι πιστεύουν οι, ε, ε κάποιοι άνθρωποι. Χρειαζόμαστε πολύ καλύτερη συνεργασία μεταξύ των βέλτιστων, των ε, ε, ε, εκείνων που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Αυτό είναι λοιπόν θα μπορεί να είναι η εδαφική συνεργασία. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση από αυτού. Πρέπει να παραμείνουμε στα 5% ως ποσοστό. Και είναι σημαντικό και για αυτά που είπε ο Γιάνν Όλμπριχτ και αναφέρθηκαν και προηγούμενα. Αν θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι, προπομπή σε αυτή την ε, προσέγγιση για τη συνεργασία για μείζονες τομείς ε, για την μακροπεριφερειακή στρατηγική που θα ακολουθηθεί για τις μακροπεριφέρειες αυτά όλα θα πρέπει να μπορέσουν να κινητοποιηθούν μέσω αυτή της κάτω προς τα άνω προσέγγισης της συμμετοχής και συνεργασίας σε αυτό το μείζον πλαίσιο μεταξύ των χωρών μας, των κρατών μας. Είδαμε καμιά φορά πρωτοβουλίες όπως για τη Βαλτική για παράδειγμα δεν κινητοποιούνται από την περιφερειακή, πολιτική περιφερειακή ανάπτυξη ή το περιβάλλον. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να παραμένουμε μέσα σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μέσω των μέσων των κανονισμών μας και γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το 5%. Να μην το απεμπολίσουμε αυτό, να μην το εγκαταλείψουμε, γιατί διαφορετικά θα σας πω τι θα συμβεί. Σε 15 χρόνια τι θα έχουμε. Θα έχουμε 15 μακροπεριφέρειες, εντάξει. Και τι θα γίνεται με αυτές θα συνεργάζονται οι χώρες ε, για αυτές και θα λένε δεν χρειαζόμαστε πλέον περιφερειακή πολιτική, πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης διότι συνεισφέρουμε ήδη για την ανάπτυξη των μακροπεριφερειών μας με αυτόν τον τρόπο. Γιατί από πλευράς ενός κράτους να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέσο για να υπάρξει ενίσχυση πόλεων ε, ή άλλων δράσεων. Λοιπόν, αυτή με την οτροπία πολλών, ίσως έστω και στην Ολλανδία. Ωραία για, το για την περιφερειακή πολιτική. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα συνεισφέρουν όμως τότε σε 15 χρόνια οι χώρες για τις μακροπεριφέρειες. Και αυτό δεν είναι καλό. Θα είναι πολύ αρνητική εξέλιξη. Λοιπόν, παραμένουμε στο 5%. Θα δώσουμε μάχη για το 5% και θα έχουμε μια πάγια ισχυρή βάση για την επικουρικότητα και για την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματο στην Ευρώπη. Αυτή είναι ακριβώ η περιφερειακή διάσταση. Ευχαριστούμε. Δεν νομίζω ότι θέλει κανεί άλλο το λόγο. Επομένω, δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Καταρχά, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία την οποία κάνει. Ο κανονισμό τη είναι πάρα πολύ τεχνικό, πολύπλοκο και πραγματικά απαιτεί να δούμε πολύ λεπτομερώς κάποια ζητήματα, γιατί κάποιες μικρές αλλαγές μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα προγράμματα. Έχουμε δει δύο βασικές προκλήσεις ουσιαστικά και νομίζω να φέρθηκε σε αυτές και η συγγήτρια. Πρώτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε ευθυγράμμιση με τον κανονισμό κοινών διατάξεων και δεύτερον, να γίνει μια διασύνδεση όσον αφορά τη συνεργασία με τα εξωτερικά μέσα. Πολύπλοκη συζήτηση αυτή στο Συμβούλιο και περιμένουμε ότι θα είναι πολύπλοκη συζήτηση και εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως να αντιμετωπίσουμε σωστά και τα δύο ζητήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όπου υπάρχουν διαφορετικά μέσα, το IPA, το Μηχανισμό Προταξιακής Βοήθειας ή τα άλλα, είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε τον κατάλληλο ευθυγραμμισμό. Διαφορετικά τα πράγματα γίνονται αρκετά προβληματικά. Όσον αφορά τώρα την μακροπεριφερειακή στρατηγική, η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν θα πρέπει να προβλεφθούν νέα κονδύλια για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Οι στρατηγικές αυτές είναι ένα μέσο συνεργασία εθελούσιο, όπου κράτη-μέλη και περιφέρειες ε, συνεργάζονται για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, και αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, τα υφιστάμενα μέσα, προγράμματα mainstream, κρατικά και διασυνοριακά, θα πρέπει να κινητοποιηθούν για τα ζητήματα τα μακροπεριφερειακά αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρα, από διαφορετικές προτεραιότητες που υπάρχουν σε χώρες και περιφέρειες. Για να στηρίξουμε λοιπόν τα μακροπεριφερειακά προγράμματα και τη μακροπεριφερειακή στρατηγική, χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτική συνοχής. Και συμφωνώ με αυτό που είπε η Επιτροπή σα, ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε καλή μακροπεριφερειακή στρατηγική είναι να εξασφαλίσουμε πολύ καλά κονδύλια στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχή και στα πλαίσια του ETC. Ευχαριστούμε, Ρίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω και όλους ε, όσοι πήραν το λόγο και κάνανε πολύ επικοδομητικά σχόλια. Να ευχαριστήσω επίσης και τους σκιώδεις συγητές, καθώς επίσης και όλους όσοι ε, συνεργάστηκαν για τις διαπραγματεύσεις τις οποίες κάναμε. Να ευχαριστήσω βέβαια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για τον κανονισμό αυτό. Όσον αφορά τον προπολογισμό, συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν από τους συναδέλφους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δική μας Επιτροπή σαφώς υπερψήφισαν το 7% για τον προπολογισμό για τα προγράμματα ETC. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εμείνουμε στα στοιχεία αυτά, να χρηματοδοτήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και να ευχαριστήσω επίσης και τον Λάμπερ, το οποίο υποστηρίζει τον προπολογισμό αυτό για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Ακούσαμε τα βασικά επιχειρήματα που δικαιολογούν αυτή τη χρηματοδότηση και συμφωνώ βέβαια. Τώρα, όσον αφορά τι περικοπέ του προπολογισμού, έχω την εντύπωση ότι η περιφερειακή συνεργασία πραγματικά θα πληγεί αν γίνει μια τέτοια μείωση. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ένα ενιαίο μέτωπο για το ζήτημα το χρηματοδοτικό. Γιατί ε, καταλαβαίνετε ότι η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί πραγματική προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά τις μακροπεριφέρειες Άρθρο δηλαδή 7 όπου προβλέπονται κοινέ ε, δράσεις. Πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής μας μετά την ψηφοφορία. Θεωρούμε ότι οι μακροπεριφέρειες δεν θα πρέπει να έχουν έναν συγκεκριμένο προπολογισμό, ξεχωριστό προπολογισμό. Θα πρέπει να ενταχθούν στο εφιστάμενο πλαίσιο ως υποκατηγορία της προβλεπόμενης περιφερειακής συνεργασίας. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σημείο αυτό. Τώρα, αν δούμε την διατύπωση του άρθρου 7, την οποία επεξεργαζόμαστε αστικά και με το Συμβούλιο, συμφωνώ ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Και ουσιαστικά κάνω μια έκκληση προκειμένου η μακροπεριφερειακή συνεργασία να αποτελεί τμήμα της περιφερειακής συνεργασίας, αλλά όπως σας είπα, όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους δεν θα πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστή χρηματοδότηση για τη μακροπεριφερειακή στρατηγική. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και στην επόμενη συνεδρίασή μας. Like the... Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε στο 14 τώρα και να μας πείτε τα σχετικά για αυτό το σημείο. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν καινούρια πράγματα, αλλά αναφέρατε το παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσω στα γερμανικά μετά από τον πολωνικό χαιρετισμό. Μετά από την Κυπριακή Προεδρία, που δυστυχώς δεν προχωρήσαμε πολύ, με τον κανονισμό αυτόν σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας. Ήρθαμε ήδη σε επαφή πέρσι με τους εκπροσώπους της ε, επερχόμενης ε, Ιρλανδικής Προεδρίας και τελείως διαφορετικός άνεμος πνέει πλέον εδώ. Ακούσαμε χθε και τον Ιρλανδό Υπουργό που είπε τον ε, Φεβρουάριο θα προσπαθήσουν στο Συμβούλιο να υπάρξει μια συνεννόηση, μια συμφωνία για τον κανονισμό ευρωπαϊκό αυτό κανονισμό για την εδαφική συνεργασία. Είχα ευκαιρία μαζί του και με τους συνεργάτες του να συζητήσω κάποια πράγματα πράγματα και μεταξύ και το Συμβούλιο στο επίπεδο εργασίας εξοικειώθηκε με τον κανονισμό εδαφικής συνεργασίας. Έχω άτυπα κάποιες πληροφορίες που μου έχουν διατεθεί επικεντρώνονται στο Συμβούλιο επί τίνος πράγματος. Οι συζητήσεις εστιάζονται σε αυτό το οποίο υποθέταμε κιόλας, ιδιαίτερα δηλαδή στο σημείο έγκρισης και το ποια διορία θα ισχύει, ποια προθεσμία θα ισχύει. Έξι μήνες λένε κάποιοι, άλλοι λένε όχι. Θα δούμε τώρα. Έξι μήνες ε, για την ε, αδειοδότηση θα πρέπει να επαρκεί ως χρόνος ε, για την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή να τοποθετηθεί. Δεν πρέπει λιγμοί να επιτραπούν ώστε τεχνητά να παραταθεί αυτή η προθεσμία περαιτέρω και από τις διάφορες περιφέρειες βλέπω ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που, με το οποίο προσεγγίζουν αυτόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την εδαφική συνεργασία, ώστε οι διαμεθοριακές, οι μεθοριακές περιοχές να έχουν δυνατότητες να δράσουν και το βλέπουν ως το κατάλληλο μέσο με το οποίο θα μπορέσουν να δράσουν και να διαμορφώσουν τις συνεργασίες τους μέσα στο πλαίσιο αυτό. Τα θέματα λοιπόν της αίγκρισης και αδειοδότησης είναι το ένα. Το άλλο, από επιμέρους τοποθετήσεις μελών του Συμβουλίου θα έλεγα, ακούγεται, δημιουργείται η υπόνοια, έστω και στο περιθώριο κάποια υποψία, ότι μέσω του κανονισμού για την ε, ε, εδαφική συνεργασία κάποιες ε, αρμοδιότητες αναδιαμορφωθούν σε σχέση με τις περιφέρειες αυτές, τις συνολικές περιφέρειες. Μπορούμε να άρουμε αυτή την υποψία. Υπάρχουν κράτη τα οποία είτε έχουν ιδιαίτερα κρατικά σχεδιαζόμενη πολιτική ή άλλα κράτη που δεν έχουν καθόλου τέτοια εδαφική προοπτική, εδαφική συνεργασίας από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου, τουλάχιστον από τα όσα μου διαβιβάστηκαν, αν ένα κράτος μέλος ή στη δική του επικράτεια ιδρύεται μια τέτοια ε, πρωτοβουλία, τότε θα μπορεί με μεθοριακές περιοχές χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει μια διασύνδεση ώστε να μπορούν δύο κράτη ας πούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο και να λειτουργούν σε αυτή τη δυνατότητα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς ε, και να το δει. Δεν είναι ανυπέρβλητα τα εμπόδια ή ε, τα προβλήματα που τίθενται και από τον Υπουργό, ε, Ιρλανδό Υπουργό όπως τα ανέφερε χθε ότι θα εγγραφεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη του Φεβρουαρίου για το Συμβούλιο για να καταλήξουν σε μια λήψη απόφασης. Έχουν κανονιστεί οι δύο διάλογοι για το Μάρτιο και ευελπιστούμε λοιπόν έτσι ότι αυτός ο κανονισμός θα προαχθεί και ότι κατά το πρώτο εξάμεινο του 2013 θα μπορέσει να ευδοκιμήσει και να ολοκληρωθεί. Μια και εδώ δεν έχουμε προβλήματα πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων, δεν πρόκειται για κονδύλια που θα επιμεριστούν, αλλά για ένα νομικό μέσο. Και έτσι λοιπόν ανεξάρτητα από τι διαπραγματεύσεις για τα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια θα μπορέσει έτσι να ρυθμιστεί. Αυτό ευελπιστούμε θα γίνει. Εν πάση συντομία αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ah. ερωτήσει, δεν βλέπω να υπάρχουν. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής από, αυτού του θέματος. Ποια είναι η άποψή σας. Όπως είπε και ο εισηγητής, ε, η Προεδρία κάνει προσπάθεια να ολοκληρώσει τις συζητήσεις του κανονισμού το Συμβούλιο για να αποκτήσει εντολή διαπραγμάτευση. Μπορούν νομίζω να το κάνουν Φεβρουάριο νομίζουμε και μετά μπορούν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Αλλά είναι τεχνικός ο τομέας. Θα απαιτηθεί αρκετό χρόνος για τη συζήτηση. Ωστόσο, αν υπάρχει ο χρόνος μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος για να ευθυγραμμιστεί χρονικά και με τα άλλα τμήματα του πακέτου. Δεν βλέπω κάποιον από την Ιρλανδική Προεδρία, δεν ξέρω κάποιο από το Συμβούλιο. Αν κάποιο από το Συμβούλιο θέλει να κάνει ένα σχόλιο, παρακαλώ. Αλλιώ εμπιστευόμαστε ότι η Επιτροπή ε, μα λέει τα σωστά πράγματα. Λαμπέρ. Επειδή τελειώνουμε τις συζητήσεις για όλα τα ζητήματα που είναι διαπραγμάτευση. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με τις δυνατότητες να πάμε στην Ολομέλεια. Τα πάντα βεβαίως εξαρτώνται εν τέλει από το δημοσιονομικό πλαίσιο. Μπορείς, ωστόσο, μπορείτε ωστόσο πρόεδρε, να μας ενημερώσετε πώς θα προχωρήσει η βάση της εντολής διαπραγμάτευσης είναι, ε, έχει μπλοκάρει το θέμα του να πάνε στην Ολομέλεια για όλα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Ακούμε για θετικές ε, προσεγγίσεις για πιθανές συμφωνίες αλλά πώς θα προχωρήσει εμείς δεν έχουμε πει να πάμε στην Ολομέλεια ποια είναι τα επόμενα βήματα η κατάσταση έχει ως εξής. Υπάρχει απόφαση από πέρσι το καλοκαίρι της διάσκεψης των πρόεδρων, όπου είχε εξηγηθεί σαφές ότι οι επιτροπές δεν μπορούν να πάνε στην Ολομέλεια πριν την έγκριση από το Κοινοβούλιο της γνωμοδότησης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η προσέγγιση μας είναι να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και όταν ανακύψει η δυνατότητα να πάμε στην Ολομέλεια να το κάνουμε. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσουν οι διαπραγματεύσει. Χθε ακούσαμε την Προεδρία που είπε ότι είναι αισιόδοξη πω θα υπάρξει απόφαση του Συμβουλίου 7-8 ε, Φεβρουαρίου. Και η εντολή διαπραγμάτευσης με το Κοινοβούλιο μάλλον ε, θα ληφθεί. Από ό,τι καταλαβαίνω η προετοιμασία του κανονισμού για το, των κανονισμών για, τα δημοσιονομικά, για τις δημοσιονομικές προοπτικές μπορεί να πάρει χρόνο. Άρα κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο τον τέλη Φεβρουαρίου. Μπορεί να κρατήσουν ένα μήνα παραπάνω. με τις διαδικασίε θα πάμε στην Ολομέλεια για το MFF. Αν έχουμε πλειοψη... απόλυτη πλειοψηφία αποφασίζουμε για το MFF. Ταυτόχρονα θα διαπραγματευόμαστε μόλις τελειώσουμε τις διαπραγματεύσεις ερχόμαστε στην Επιτροπή για να έχουμε την έγκριση της Επιτροπής και κατόπιν πηγαίνουμε στην Ολομέλεια. Δεν περιμένω να υπάρξει οποιαδήποτε παρεμπόδιση της δυνατότητας να πηγαίνουν οι επιμέρους επιτροπές στην Ολομέλεια ξεχωριστά με τους κανονισμούς. Δεν νομίζω ότι η ιδέα είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθούν και 60 κανονισμοί γιατί αυτό θα είναι παράλογο και θα μπλοκάρει όλη τη δουλειά στο Κοινοβούλιο. Ε, πιστεύω ότι όταν είμαστε έτοιμοι θα πάμε στην Ολομέλεια και ανάλογα με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί αν θα πάμε για την ε, πρώτη ανάγνωση ή για μόνη ανάγνωση. Αυτό από εμάς εξαρτηθεί. Και από εμάς εξαρτηθεί επίσης αν θα πάμε με ένα, με ένα ενιαίο πακέτο ή όχι. Ή αν εάν είμαστε έτοιμοι με το γενικό κανονισμό θα πάμε πρώτα με αυτόν. Μαζί θα το αποφασίσουμε. Πάντως δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ενιαία θέση των αρχών των, του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το πώς θα προχωρήσουμε προς την Ολομέλεια. Αυτά. Και αυτά θα πω και ως θέσεις της Επιτροπής σε οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση υγιεινή μέχρι το επίπεδο του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι και οι υπηρεσίε ε, την ίδια θέση είχαν. Όταν είμαστε έτοιμοι, πάμε στην Ολομέλεια. Συμφωνώ. Το καταλαβαίνω. Ο στόχος είναι να έχουμε αποτελέσματα. Άκουσα ότι άλλες επιτροπές θα πάνε για εντολή στην Ολομέλεια. Δηλαδή ψήφισε η Γεωργική Επιτροπή και μετά θα πάνε στην Ολομέλεια για, για εντολή με πλήρη συζήτηση. Εμείς άλλη γραμμή ακολουθούμε. Αλλά οι προσπάθειές μας θα έπρεπε να είναι ορατές και στην Ολομέλεια όποτε είναι δυνατό. Νομίζω ότι κάνουμε πολύ πρόοδο Ακούω ωστόσο από εδώ και από εκεί συναδέλφους που λένε ότι την άλλη φορά μπορεί να είστε ε, εκδημοκρατισμός, ε, τι θα κάνουμε με την επόμενη ε, Επιτροπή μετά το 16 δεν καταλαβαίνουν ότι εμείς ετοιμάζουμε μία πολιτική για τα επόμενα 6 χρόνια. Αν δεν φέρουμε το θέμα μπροστά για συζήτηση, δίνουμε τη δυνατότητα σε άλλους να λένε αυτό είναι ένα ασήμαντο κομμάτι του προπολογισμού, το αφήσουμε για μετά. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ενημέρωση είναι χρήσιμη και εξετάστε το πότε να πάμε στην Ρωμέλεια. Να σας πω επίσης κάτι που δεν είπα. Το είπα όμως χθες στους συντονιστές. Οι συνάδελφοι που έχουν δικές τους εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλία. θα έπρεπε να έχουν μια πολιτική για το πώς θα πηγαίνουν πότε θα πηγαίνουν στην Ολομέλεια, να έχουμε μια συζήτηση ας πούμε στο Στρασβούργο για θέματα πολιτικής, ε, αν κλείνουμε γρήγορα αυτά που, που είναι κρεμή τώρα, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα παρουσιάζουμε. Και γενικά καλό θα ήταν να τελειώνουμε με τις εκθέσεις που έχουμε να λάβει πριν το τέλος της φοιτίας μας. Με αυτά θα κλείσω αυτό το πακέτο της συνάντησης. Έχουμε μια, ένα νέο σχέδιο, ένα ακόμα σχέδιο γνωμοδότησης. Χωακίμ δεν σου έδωσε το λόγο. Τον ζήτησε. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα μόνο αυτό το οποίο είπε ο Λάμπερτ ε, να δούμε και να το υποστηρίξω και πάλι αυτό. Εμείς δηλαδή κάπου σε ένα ενδιάμεσο βήμα που θα κάνουμε να περάσουμε στην Ολομέλεια με αυτό. Επειδή ακούω και επίσης από πολλούς συναδέλφους ε, που δεν ε, ε, ε, έχουν εμβαθύνει τόσο στα θέματα της διαθωτικής πολιτικής με ρωτάνε τι γίνεται με εσά για αυτό το θέμα να συζήτηση στην Επιτροπή Γεωργίας ή στην Επιτροπή Αλίας εν τω μεταξύ γίνεται πόλεμος μεσαιωνικός εκεί μεταξύ των μελών και υπάρχει κάποια ανησυχία ότι χωρίς κανένα θόρυβο και φασαρία προχωρούμε εμείς. Ρωτάνε τι κάνετε εσείς αν έχουμε ένα δεδομένο αποτέλεσμα και πάμε στην Ολομέλεια από πλευρά μας και πούμε ότι ή θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί, ε, τότε ίσως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε συζητήσεις που θα ήταν περιτές. Γιατί για την ε, πολιτική συνοχή ε, έχουμε 40% της, των κονδυλίων της πολιτικής μας. Και πιο πριν το να πάμε στην Ολομέλεια θα έπρεπε να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουν κάποιες πληροφορίες οι συνάδελφοι γι' αυτό και να πούνε εντάξει ωραία διαπραγματεύεστε σωστά για αυτό το θέμα θέμα. Τώρα ολοκληρώστε το σχετικά. Ευχαριστώ. Well, as you know, ε, όπως γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε Χωακίν, έχουμε ένα ειδικό μέσο, μια ειδική ξεχωριστή πλατφόρμα την οποία την αποκαλούμε Working Party, ομάδα εργασίας για τη μελλοντική πολιτική σχετικά και λόγω των διαπραγματεύσεων έχει προσκληθεί και επανειλημμένα και για τα θέματα απασχόλησης. Είχαμε μια συνάντηση όπου προσκαλέσαμε και τους εισηγητές των άλλων εμπλεκόμενων πέντε ταμείων των Ευρωπαϊκών Διαθωτικών Ταμείων και επενδυτικών ταμείων. Έχουμε και την ανταλλαγή επιστολών, ιδιαίτερα με την κυρία Μπέρες και έτσι υπάρχει ας το πω έτσι η πρόθεση νομίζω από πλευράς μας να τους εξοικειώσουμε και να συνειδητοποιήσουν, ε, να ευαισθητοποιηθούν περί τίνος πρόκειται. Ένα πράγμα είναι η συνεργασία με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές και άλλο πράγμα είναι το θέμα της Ολομέλειας. Δύσκολη επιλογή θα είναι. Όταν θα έχουμε 85 ε, ή 90% του ε, γενικού κανονισμού που θα έχουμε ολοκληρώσει και θα έχουμε καλύψει, τότε μπορούμε να δούμε μια τέτοια δυνατότητα. Αλλά ας περιμένουμε και ας το δούμε μετά. Ας κάνουμε πρώτα τη δουλειά μας, να διαπραγματευτούμε αποτελεσματικά όσο πιο γοργά γίνεται και ας αναμείνουμε την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής και ας δούμε μετά ποια θα είναι η θέση του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτό και θα λάβουμε σχετικά απόφαση πώς θα προχωρήσουμε με αυτό. Δεν θέλω να συνεχίσουμε με κάποιες εικασίες τώρα εδώ και να πιθανολογούμε το ένα ή άλλο θα πρέπει να επιλέξουμε και να δούμε στη συνέχεια. Θα πάμε για την πρώτη ανάγνωση ή σε μία ανάγνωση θα ολοκληρώσουμε ή θα έχουμε πρώτη και δεύτερη. Άλλο, όλα αυτά θα επηρεάσουν τα πράγματα και θα δούμε πώς θα προσεγγίσουμε το θέμα της ψήφισης στην Ολομέλεια. Θα συνεχίσουμε όμως και τη συζήτηση επ' αυτού με τους συντονιστές επίσης. Να πω και πάλι, ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Τέτσεβα θα έρθει πιο νωρίς για αυτό το ένα σημείο και θα είναι σύντομο ελπίζω σε 15 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε με αυτό το σημείο για εκείνη ε, η Ρίκα τώρα σε σχέση με τη γνωμοδότηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην αγορά παρακαλώ σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να αναφέρω το εξής πρώτα απ' όλα βέβαια θα είμαι σύντομη Ωραία. Είναι μια γνωμοδότηση λοιπόν αυτή για τις ε, πηγές ανανεώσιμες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προκλήσεις και ευκαιρίες ε, που προσφέρονται από αυτή την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από κοινού και με την επί της ουσίας αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ήτρε παίρνουν ιδιαίτερα σοβαρά αυτή την πτυχή των ανανεώσιμων οι πολίτες ε, και υπό το πρίσμα της Περιφερειακής Επιτροπής εξετάζουμε λόγω διαφορετικών περιοχών και περιφερειών της Ευρώπης μια και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα δίνει ευκαιρίες εκεί στις περιφέρειες της Ευρώπης να δραχθούν της ε, προοπτικής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπάρχουν λοιπόν ευκαιρίες και τα, στο μέλλον, τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε. Θέλω να υπογραμμίσω το θέμα της χρηματοδότησης. Είναι σημαντικό νομίζω αυτό και για τα μέσα και διευκολύνσεις ε, του Ταμείου Συνοχής που όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε για να επικεντρωθούν τα κονδύλια στις επενδύσεις δηλαδή που θα γίνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή είναι η σωστή πορεία προς το μέλλον για να διασφαλίσουμε την πτυχή της ανα... ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μας ε, αυτή η χρηματοδότηση, αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα και διευκολύνσεις να μπορέσουν να δράσουν ε, στοχευμένα και από κοινού και με τη στόχευση του ορίζοντα 2020 και της στρατηγικής ε, μέχρι το 2020. Ξεκινώντας από κάτω-κάτω, εκ των κάτω προς τα άνω, έχουν γίνει έρευνες ε, για την περιφερική ανάπτυξη και για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ανάπτυξης πηγών ενέργειας για αυτή την περιφερειακή ανάπτυξη. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να υπάρξουν βελτιώσεις όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό μέσω του προγράμματος Ελένα προγράμματος αρρωγήσια και ενίσχυσης και για την ε, ανάπτυξη συγκεκριμένα και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ε, σε σχέση με τα θέματα ενέργειας χρησιμοποιώντας αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει σε αυτόν τον τομέα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την αυτάρκεια όσον αφορά τα ενεργειακά προϊόντα. Να δώσουμε ένα σημαντικό δηλαδή ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μπορέσει να προσεγγιστεί και να επιτευχθεί η αυτάρκεια. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή πιο αποτελεσματικά ευρωπαϊκές πηγές ενέργειας αντί να εισάγουμε, εισαγάγουμε άνθρακα ή ορυκτά αλλά καύσιμα από την αλλοδαπή. Του, του λεχθέντος τώρα πιστεύω ότι θα έπρεπε να στρέψουμε ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιομορφίες και ανάγκες ξεχωριστές της κάθε ευρωπαϊκής περιφέρειας δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια ισοπεδωτικά πολιτική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για όλες τις συλλήβδιν τις περιφέρειες της Ευρώπης. Σε διασύνδεση με αυτό θα ήθελα να πω πόσο σημαντικά είναι τα θέματα της, βιο, ε, των, της βιοενέργειας. Για παράδειγμα, να δώσουμε μια νέα προώθηση στις γεωργικές περιοχές και τις περιοχές της υπαίθρου με τα βιοπαραγόμενα. Επίσης, σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και σε ένα άλλο θέμα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ένα διασυνοριακό σκηνικό, διαμεθοριακά. Και αυτό μας εντάσσει στο πρόγραμμα όσον αφορά το σχέδιο της ε, Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης. Ε, θα βοηθούσε λοιπόν η διασυνοριακή συνεργασία και συνιστόσα. Τα επόμενα χρόνια έχουμε αρκετές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη. Αν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και ε, είμαστε στεφτοί με επιτυχία το εγχείρημά μας για την, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μακροπρόθεσμα στεφθούν με επιτυχία οι προσπάθειές μας. Πρέπει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο στην αηφορία να το δούμε, στην βιωσιμότητα. Έχουμε μια αντιφατική πολιτική για τα θέματα ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Έχουμε διαφορετικούς στόχους ε, που θέλουμε να επιτύχουμε, όμως από πλευράς ε, περιβαλλοντικών δράσεων θέλουμε κάποιες ε, πηγές από αυτές τις δράσεις να μειώσουν για παράδειγμα τις εκπομπές ρήπων και τα λοιπά. Θα πρέπει διασυνοριακά και συν, ε, οικουμενικά σφαιρικά να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές σε τέτοια ενεργειακά θέματα. Θέλουμε να αναφέρουμε αυτά τα θέματα σε αυτή τη γνωμοδότηση. Προσβλέπω στα σχόλια παρατηρήσεις σας για αυτή τη γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ποιος αντικαθιστά το Μάρκους Πίπερ, εσύ Λάμπερτ μάλιστα, έχεις το λόγο λοιπόν. Ο Μάρκος είναι αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Βιομηχανίας. και ουσιαστικά εργάζεται για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα, για την έκθεση αυτή. Δυστυχώς δεν μπορεί όμως να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Μου είπε πάντως ότι το σχέδιο αυτογνωμοδότησης είναι πολύ καλό. Και είπε επίσης ότι θα πρέπει πραγματικά να δούμε ποιε δυνατότητε συμπληρωματικότητα υπάρχουν στα διάφορα εφιστάμενα μέσα. Βέβαια, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική από χώρα σε χώρα και εντελώς διαφορετικές επιλογές τεχνολογίας γίνονται τελικά από τη μία περιφέρεια στην άλλη, από τη μία χώρα στην άλλη. Από την άλλη όμως, πρέπει κανείς να σκεφτεί και το ζήτημα του κόστου ωφέλου, της αποδοτικότητας. Αναφέρθηκες και εσύ στο ζήτημα αυτό. Ενδεχομένω κάποιο να θέλει να πτύξει περισσότερο την ηλιακή ενέργεια στη Φιλανδία. Ωστόσο όμως θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δει κανείς αν κάτι τέτοιο θα ήταν ε, οικονομικά αποδοτικό, αν ε, υπάρχει λόγος για μια τέτοια επένδυση. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Γερμανίας. Και ας δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, στους πολίτες. Το ζήτημα της οικονομικής αποδεκτικότητας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί πραγματικά να επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή των πολιτών. Και αυτό συνδέεται επίσης και με την Στρατηγική Ευρώπη 2020. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι που κάνουμε εδώ πέρα για την ενέργεια θα μπορούν ουσιαστικά να αναλυφθούν οικονομικά από τους πολίτες, ότι θα τους βαρύνουν πάρα πολύ. Και μία σχετική τροπολογία θα ήθελα να υποβάλω. Και έπειτα υπάρχει και το ζήτημα της σχέσης της πρότασης αυτής με τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Ξέρετε ότι η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την αιωλική ενέργεια και τις σχετικές τεχνολογίες. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να εκχωρήσουμε μέρος της δικής μας τεχνολογίας σε άλλες τρίτες χώρες, για παράδειγμα τις χώρες της Ασίας. Έχουμε κάποια πολύ καλά προγράμματα, τον ορίζοντα 2020 και αναφέρθηκε σε, σε αυτά στην γνωμοδότησή του. Τώρα όσον αφορά τα ευφυή δίκτυα ενέργειας, τα smart grids. Γι' αυτά προβλέπεται ένας υψηλός βαθμός αποκέντρωσης. Τα προβλεπόμενα πάντως δίκτυα δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν μπορούν να πάρουν το πλεόνασμα ενέργειας που υπάρχει σε μία περιφέρεια και να το μεταφέρουν σε μία άλλη. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές στις κάτω χώρες ενδεχομένως να έχουμε ένα απόθεμα, ένα πλεόνασμα αιωλικής ενέργειας σε μία περιοχή, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε σε μία άλλη περιοχή που θα μπορούσε να το αξιοποιήσει. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα και θα πρέπει να εκπονήσουμε ένα σύστημα που θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Πολλές φορές ασκείται τόση πολλή πίεση, υπάρχει τόση μεγάλη ζήτηση από το ενεργειακό δίκτυο μιας περιοχής που το δίκτυο καταραίει. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε όχι σαν απειλή, να το εξετάσουμε περισσότερο σε ευκαιρία για περισσότερες επενδύσεις και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ενδεχομένως να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποια smart grids, τα οποία θα λειτουργούν αποτελεσματικά με ένα σύστημα αποκέντρωσης που θα μπορούν εύκολα να μεταφέρουν με ενέργειες από τη μία περιοχή στην άλλη. Τα εφή δίκτυα χρησιμοποιούν τεχνολογία που στηρίζεται στην πληροφορική, στην ε, διαχείριση πόρων και ξέρετε ότι στην ε, έκθεση της κυρίας Κολάρσκα Μπαμπίνσκα γίνεται αναφορά σε αυτές τις ε, ευκαιρίες. Το ζήτημα λοιπόν το έχουμε συζητήσει εκτενώς και στην προηγούμενη μας συνεδρίαση. Συγχαρητήρια πάντως για την γνωμοδότησή σου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σταυρακάκης έχει το λόγο που αντικαθιστά τη Μαρία Ριγκόγιν. Κύριε Πρόεδρε, η συνάδελφός μας ε, Μαρία Ριγκόγιν Πέρες δεν μπορεί να βρίσκεται σήμερα μαζί μας καθώς βρίσκεται στη Χιλή συμμετέχοντας στις ενέργειες της κοινή κοινοβουλευτική Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής και της έκτης Συνόδου Ρωμέλειας της Eurolat. Για τον λόγο αυτό μου ζήτησε να μεταφέρω τις θέσεις της σχετικά με το σχέδιο γνωμοδότησης τη κυρία Ρίκα Μάνερ για τι σημερινέ προκλήσεις και ευκαιρίε για την ανανεώσιμη ενέργεια. Πρώτα απ' όλα εκ μέρου τη κυρία ε, Ιργκόγεν Πέρες, αλλά και προσωπικά θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μάνερ για την εξαιρετική τη δουλειά. όπω έχει επισημάνει η συγγήτρια, η ανανεώσιμη ενέργεια βελτιώνει την οικονομική ανάπτυξη και τι εξαγωγικέ ευκαιρίες των περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντα νέε βιομηχανίε και καινοτομία, και αυξάνοντα επίση τον αριθμό των θέσεων εργασία, ιδιαίτερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Επιπλέον, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια συμβάλλουν στην ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, στην διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού τη Ευρώπη και στην ενεργειακή αυτάρκεια. Δεύτερον, η πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση και να δώσει ισχυρή έμφαση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία για τον λόγο αυτό η πολιτική συνοχή χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ένα κατάλληλο και παρκή προπολογισμό για την περίοδο 2014-2020. Τρίτον, οι περιφέρειε τη Ευρώπη θα πρέπει να έχουν αρκετή ευελιξία για να επικεντρωθούν σε αυτέ τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, οι οποίε είναι οι κατάλληλε για τι τοπικέ του συνθήκε, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2020 και για μια βιώσιμη και καθαρή ανανεώσιμη ενεργειακή οικονομία μέχρι το 2050. Τέλος, η κυρία Ιρικόγεν Περές θα ήθελε να υπογραμμίσει τη σημασία της αύξησης του αριθμού και της βελτίωσης των διασυνοριακών συνδέσεων που αποτελεί ζήτημα ύψης της σημασίας για την επιτυχία της ενιαίας αγοράς και την ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης προτείνει η ενίσχυση από το πρόγραμμα Ελένα να υποστηρίζει πιο αποτελεσματικά μεγάλης κλίμακας επενδυτικά σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης το πρόγραμμα Intelligent Energy η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει περαιτέρω την αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με βάση όλα αυτά τα σχόλια, η κυρία Ειρηγόγεν Πέρε προτίθεται να καταθέσει εκ μέρου τη πολιτική ομάδα του SD ορισμένε τροπολογίε για να ενισχυθούν ορισμένα συγκεκριμένα σημεία τη ε, νομοδότησή σα. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταυρακάκη. Δεν ξέρω, θέλει κάποιος από τους πράσινους να λάβει τον λόγο, όχι. Μια στιγμή. Φρανσουά Αλφονσί, εσείς. Οκ, πάτε πάρτε τον λόγο παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Ζακομπή που είναι ο υπεύθυνο ε, μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονοματός του για να υπογραμμίσω το πόσο ενδιαφέρουσα είναι η έκθεση αυτή στην παρούσα φάση όταν υπάρχει μια στρέβλωση μεταξύ των στόχων που έχει θέσει η Ένωση και της πραγματικότητας που βλέπουμε επιτέπου ιδιαίτερα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια που διέρχεται μια κρίση που, επιτρέπει, που δεν μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε στην, ε, στους στόχους μας αν δεν λυθεί η κρίση. Η ομάδα μας, η οικολογική ομάδα, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις υποδομές ε, των ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργεια και συμφωνώ με, απόλυτα με αυτό που είπε ο Λάμπερτ για τις επενδύσεις στο δίκτυο που πρέπει να γίνουν ουσιαστικοί προτεραιότητα για να αυξηθεί η εμπλοκή των νεώσιμων πηγών ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Παραμένει ένα σημαντικό δυναμικό που δεν έχει τύχη εκμετάλλευση και απαιτεί επενδύσεις. Επενδύσεις κυρίως από τον δημόσιο κορβανά, ιδιαίτερα δε από την Ευρώπη. Η σύγχρηματοδότηση και ο ιδιωτικό τομέα προφανώς πρέπει να συμβάλλουν για να αλλά πρέπει πρώτα να δώσουμε ασφάλεια και η ασφάλεια παρέχεται από δημόσιους πόρους, ιδίως από τις ένωσης, ε, πόρους Ένωσης για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, το, το υπογραμμίζω αυτό, την κρίση που ε, διανύουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η προσέγγιση της ομάδας μας. Βεβαίως είμαστε υπέρ της γνωμοδότησης και θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω το κείμενο με τις ιδέες μας, ώστε να έχει τον καλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Ευχαριστώ. Ιωχήμ. Ναι, σας ευχαριστώ. Και σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν, ευχαριστώ. Ο Λάμπερτ είπε ότι πρέπει να το διασυνδέσουμε αυτό με την έκθεση της συναδέλφου Κολάνσκα Μπομπίνσκα που στην τελευταία ολομέλεια στο Στρασβούργο την ε, ψηφίσαμε Θέλω να υπενθυμίσω ότι ακούστηκε από κάποιους συναδέλφους ότι είχαμε και μια έκθεση πριν από λίγο καιρό για τις ενεργειακές υποδομές για το 2020 ή το 2050. Και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες αυτό είναι η λιδία λίθος, αυτό είναι το φλέγον θέμα. Διαπιστώσαμε ότι για την διασφάλιση, διατήρηση του ενεργειακού δικτύου όπως υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα πόρο απέχουμε από μια, από μια ενιαία αγορά ή από μια ευρωπαϊκή διασύνδεση και χρειαζόμαστε 280 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε, να διατηρήσουμε το δίκτυο αυτό σε ένα υψηλό επίπεδο. Μια περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου θα απαιτούσε άλλα 800 δις, 800 δις. Όλα αυτά εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τότε χρησιμοποιήθηκαν ως θεμέλια για την έκθεση που συντάξαμε για τις υποδομές. Αυτά να τα δούμε λοιπόν. Δεν επαρκεί ούτε και το επόμενο Ταμείο Συνοχής για να διατεθούν αυτά τα κονδύλια. Από αλλού πρέπει να αντληθούν, άλλο μέσο πρέπει να εξευρεθεί. Το θέμα δεν είναι τώρα η υλοποίηση των στόχων 2020 που δεν μπορούν να επιτευχθούν ούτε για την παραγωγή ενέργειας. Μου λένε κάποιοι παραγωγή ενέργειας μέσω αιωλικών πάρκων για παράδειγμα, για αυτή την παραγωγή πανευρωπαϊκά οι πιθανές έδρες έχουν ήδη καθοριστεί, έχουν ήδη προσδιοριστεί για αυτά τα αιωλικά πάρκα. Η παραγωγή από τις αιωλικές αυτές ε, αντλίες έχει νόημα να γίνεται εκεί όπου είναι ισχυρός ο άνεμος, εκεί όπου είναι πολυάνεμες οι περιοχές. Τώρα, μπροστά στις ακτές, Εκεί εντωμεταξύ μέχρι και την Πολωνία θα είχαμε δυναμικό. Παντού δηλαδή έχουν προσδιοριστεί, προ-προσδιοριστεί αυτές οι έδρες, τα σημεία που θα τοποθετηθούν. Μόνο που πρέπει να μεταφέρεται η ενέργεια εκεί όπου χρειάζεται αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα. Και πάλι φτάνουμε στο ερώτημα, τι γίνεται με το δίκτυο και την επέκτασή του για να επιτευχθεί αυτό. Και είπε ο Λάμπερ, τι ζήσαμε στη Γερμανία, τι συνέβη στη Γερμανία. Η ε, επέκταση του αιτίου χρειάζεται ε, ασφάλεια σχεδιασμού, νομική βεβαιότητα και ασφάλεια. Αν υπάρξουν κάποιες αλλοιώσεις, αλλαγές ή καθυστερήσεις, για, επειδή για παράδειγμα υπάρχει κάποιο φράγμα ή κάποιο μνημείο, ε, οτιδήποτε που πρέπει να προστατευθεί και δεν μπορούν να περάσουν μεγάλοι τέτοιοι πυλώνες του δικτύου μπροστά σε κατοικημένες περιοχές κτλ. Είναι όλα αυτά θέμα κόστους. Και τι θα γίνει, θα τα πληρώσουν τα σπασμένα οι πολίτες π.χ. στη Γερμανία Γερμανία και το νιώθουν αυτό στη τσέπη τους να βαραίνει και για τους μεγάλους βιομηχανικούς τομείς που είναι ενεργοβόροι οι τιμές, ε, οι ενεργειακές πηγές ε, λένε ότι κοστίζει το ηλεκτρικό ρεύμα τόσο ακριβά, είναι τόσο δαπανηρό αυτό που θα εγκαταλείψουν την έδρα τους στην Ευρώπη, στη Γερμανία και στην Ευρώπη και θα πάνε σε άλλες χώρες όπου είναι φθηνότερη η ηλεκτρική ενέργεια. Το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο και σύνθετο. Δεν μπορούμε να το απομονώσουμε και να επικεντρωνόμαστε μόνο σε μία συνιστή τόσα ή ένα δεδομένο. Και αν δούμε τι γίνεται στη Γερμανία ή σε άλλε χώρε, ε, για παράδειγμα, σε άλλε χώρε πέρα από τη Γερμανία που συγκλονίζονται από την ε, υπερχρέωση, την κρατική υπερχρέωση, δεν βλέπουμε με ποιο τρόπο θα διατεθούν τα κονδύλια. Η φαντασία μα δεν επαρκεί για να το ε, καλύψει αυτό, για να παραμείνουμε όχι μόνο σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά και να επεκτείνουμε το δίκτυο ακόμα παραπέρα όπω θα χρειαστεί. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. και όπω ανέφερε και η Ρίκα, εκεί όπου σε αποκεντρωμένες λύσεις μπορούμε να προχωρήσουμε, να ψάξουμε να βρούμε αυτές τις λύσεις. Ο μεγάλος στόχος όμως ε, για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή ενιαία αγορά και για μια, ε, ένα δίκτυο ευρωπαϊκών χωρών για την παραγωγή ενέργειας ε, πρέπει να παραμείνει μπροστά μας, αλλά να τον διατηρήσουμε το στόχο, αλλά ο διάολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, να μην το ξεχνάμε αυτό στη συζήτηση αυτών των θεμάτων. Ευχαριστώ, εδώ. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Επίκαιρη έκθεση και έκθεση που ευθυγραμμίζεται με τις κυρίες Μπομπίνσκα αλλά και με άλλες εκθέσεις και συζητήσεις που είχαμε πρόσφατα. Ως ε, εισηγητής για το Ταμείο Συμμαχής χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη συζήτηση διότι αυτό που κάνει τώρα η Ρίκα είναι μία σαφής πρόσκληση να εγκαταλείψουμε το βραχι πρόθεσμο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. Αυτό τον ε, βραχυπροθεσμισμό που έλεγε και ο Μόντι. Έρχονται και μας λένε πάρτε ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα αλλά από την άλλη διακινδυνεύουμε να χάσουμε την ανταγωνιστικότητα για τα κράτη-μέλη, ενώ η έλλειψη ρευστότητας δεν επιτρέπει την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων. Αυτό που είναι σαφές είναι πρώτον η ανάγκη μεγαλύτερης επένδυσης στα ανανεώσιμα. Η έκθεση του 2011 λέει ότι πρώτη στη σειρά είναι η Κίνα, δεύτερη η Ευρώπη συνολικά, αλλά με μεγάλες αποκλήσεις και τρίτη είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η δεύτερη ιδέα. Όταν επενδύεις στην έρευνα και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πώς θα μπορέσουμε να παράσουμε πρόσβαση σε κοινότητες, σε περιφέρειες για τις νέες τεχνολογίες. Διότι η τεχνογνωσία είναι ακριβή οι ευρωπαϊκές εταιρείες που πηγαίνουν στην Κίνα σήμερα και δουλεύουν εκεί την παραγωγή τους στην χώρα, ξαναπουλώντας την Ευρώπη κατόπιν, γιατί είναι φτηνότερο στην Κίνα, το καταλαβαίνω, αλλά η τεχνογνωσία μας που είναι κυρίαρχη τώρα χάνεται. Μπορούμε με κάποιο τρόπο να διαφυλάξουμε την ικανότητά μας όχι μόνο να επιβραβεύουμε δημόσια το ρόλο μας αλλά να τον υλοποιούμε και στην πράξη διότι αν δούμε τα, τα γεγονότα σήμερα τη να μονάδα για παράδειγμα θα δείτε ότι δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα για την Ευρώπη αναφέρθηκε ήδη πολλοί και στη Ρουμανία ακόμα νομίζουν ότι η χρήση των ανανεώσιμων αυξάνεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, διότι αυτοί πληρώνουν μόνο τη διαφορά από την παραγωγή μέσω ρηκτών καυσίμων στην παραγωγή μέσω ε, φωτοβολταϊκών ή ανεμογεννητριών. Από την άλλη, πρέπει να αποδεχθούμε ότι η ιδιωτικοποίηση δεν ήταν πανάκια στη Ρουμανία και δεν φαντάζομαι μόνο εκεί. Βλέπουμε ότι η αύξηση, οι κορυφές της παραγωγής χειμώνα ή καλοκαίρι δίνουν μια εξαιρετικά ευέλικτη παροχή ενέργειας σε ό,τι αφορά την ένταση και το βολτάζ που δημιουργεί πρόβλημα Ξέρετε ότι αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη Ρουμανία και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους πελάτες μας. Αν ωστόσο η, Ελλάδα, η Ευρώπη συγγνώμη, θέλει να έχει μια ενοποιημένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο και όχι μόνο βραχυπρόθεσμο, γιατί το βραχυπρόθεσμο μας λέει σταθείτε στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Αυτό θα είναι εξαιρετικά θετικό για τις πολυεθνικές που μας πουλάνε πετρέλαιο και φυσικό αέριο με τεράστια κέρδη θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πελατών και τα προβλήματα των δικτύων που είναι προβληματικά, είναι παλιά, χρειάζονται ανανέωση, χρειάζεται νέες δομές αυτές που λένε τα έξυπνα δίκτυα διανομής και όλα αυτά απαιτούν τη χρήση διαρθρωτικών πόρων και πόρων συνοχής για να ελοπιδούν. Ευχαριστούμε Βίκτορ. Θέλει να απαντήσει η Επιτροπή. Παρακαλώ από την Περιφερειακή Ανάπτυξη, ε, από την κοινική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης, όχι ενέργειας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την ε, εισηγήτρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ των προτάσεων αυτών. Πρέπει πραγματικά να τονίσουμε το ρόλο που μπορούν να δραματίσουν διάφορα ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό επίση που τονίστε τη διασύνδεση με την περιφερειακή ανάπτυξη καθώ επίση και τι ενεργειακέ υποδομέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν πόρε σε περιφερειακό επίπεδο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στην Ευρώπη. Συμφωνούμε λοιπόν με όλε τι προτάσει που γίνονται. Μάλιστα, από την Γενική Διεύθυνση Ενέργεια, λοιπόν, ήσασταν. Η Ρίκα θέλει τώρα να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχολείο τη και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφου για την πολύ καλή ε, συνεισφορά από πλευρά του ε, με παρατηρήσει που μπορώ να εντάξω στη γνωμοδότησή μου. Είναι ένα πολύ σύνθετο και περίπλοκο ζήτημα αυτό το θέμα τη ε, αυτάρκεια ε, στα ενεργειακά θέματα, αλλά και των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και τη χρήση του Περίπλοκο και σύνθετο για την Ευρώπη ζήτημα. Ο Βίκτορ πραγματικά τόνισε πόσο σημαντική είναι η μακροπρόθεσμη συνιστόσα της στρατηγικής μας. Ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας είναι πολύ σημαντικό στην λήψη απόφασης αυτό εμπλεκόμενοι στις αποφάσεις από διάφορους τομείς πρέπει να γνωρίζουν πώς θα επενδυθούν αυτά τα κονδύλια σε αυτούς τους διαφορετικούς τομείς. Υπάρχουν πολλές αλλαγές, ε, ε, μεταβολές, ε, δημιουργείται αβεβαιότητα πολλές φορές όσον αφορά και καθυστερήσεις ή την δυνατότητα διευθέτησης αυτών των επενδύσεων σε σχέση με την ενεργειακή αγορά. Πρέπει λοιπόν τούτων λεχθέντων να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ενός ευρύτερου χρονορίζοντα. Το υποστηρίζω αυτό. Κάνοντας λόγο για μια γνωμοδότηση τώρα από την Επιτροπή, ε, Περιφερειακή Επιτροπή, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ποια είναι η εντολή μας. Δεν μπορούμε επί παντός του επιστητού να εντάξουμε κάθε είδους πρόταση σε μια τέτοια σύντομη γνωμοδότηση από πλευρά μας. Ο Λάμπερτ Φανίστερ Ρόι έκανε λόγο για την ε, ε, αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα κόστη και την αηφορία ε, ή την αποτελεσματικότητα γενικότερα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Η ηλιακή ενέργεια είναι σε σχέση με το κόστος πιο ευνοϊκή στην Πορτογαλία από ότι στη Φινλανδία. Λογικό αυτό, εύληπτο, πρέπει να το τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε τις ιδιαιτερότητες και το δυναμικό που έχει ξεχωριστά η κάθε περιφέρεια που μπορούμε σε αυτή να αναπτύξουμε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν σημαντικότατα θέματα τα οποία θίγονται, καλύπτονται σε αυτή τη συζήτηση και θα εντάξω αυτές τις πτυχές, αυτή τη γνωμοδότηση από κοινού με τους κοιόδης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η 28 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι Δευτέρα είναι η ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών. Λαμπέρα, θα μιλήσει μετά την εισηγήτρια. Ένα αίτημα απλώς έχω. Μπορεί να είναι στις 6 το απόγευμα η ε, καταληκτική ημερομηνία στις 28, 28 Ιανουαρίου 6 το απόγευμα για την κατάθεση τροπολογιών. Ναι, ναι, εντάξει, η γραμματεία είναι πολύ γενναιόδορη και μας επιτρέπει να πάμε μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη θητεία του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τους Ρωμά με χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αρμόδια για το πρόγραμμα αυτό. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε μέχρι το 2012 και σήμερα έχουμε την κυρία Τσαρλίνα Βιτσέβα μαζί μα, Διευθύντρια από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Ανάπτυξη, η οποία αν δεν κάνω λάθο θα μα κάνει μια παρουσίαση για την ένταξη των Ρωμά και έχει μαζί τη και κάποιους προσκεκλημένους. Κυρία Τσαρλίνα Βιτσέβα, έχετε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα είναι χαρά για μένα να παρίσταμε εδώ σήμερα. Η ομάδα μας από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά πολύ άριθμη. Έχουμε συναδέλφους όχι μόνο από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής αλλά και έχουμε και από την Υπηρεσία για την Απασχόληση και από άλλες γενικές διευθύνσεις. Προσπαθούμε πάντα να είμαστε από κοινού και να συνεργαζόμαστε όταν έχουμε θέματα που αφορούν τους Ρωμά, τους Τσιγκάνους, διότι γνωρίζουμε πόσο πολυδιάστατο είναι αυτό το πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο και πώς πρέπει και πολυδιάστατα να συνεργαστούμε για να το αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Θέλω να σας παρουσιάσω τις προοπτικές ε, περί τίνος ε, ε, επρόκειτο με αυτό το εγχείρημά μας. Ποιες ιδέες το ενέπνεαν ποια είναι τα αποτελέσματα και ποια είναι τα συμπεράσματά μας, συστάσεις τελικά. Διότι οποιοδήποτε τέτοιο ε, σχέδιο υπάρχει για να εξεταστούν και να αξιολογηθούν κάποιες δραστηριότητες, να υπάρξουν ε, συμπεράσματα που θα μπορέσουν να ενταχθούν στην κυριότερη, ευρύτερη πολιτική και θα εμπνέουν τις δραστηριότητες αυτές της δράσης αυτής της πολιτικής στη συνέχεια. Όπως είπατε Πρόεδρε ευθύ εξ αρχής, μάλιστα ελπίζω ότι όλοι είναι σε θέση να δουν τα γραφήματα, της διαφάνειες. Αυτό το ε, σχέδιο ε, δόθηκε με εντολή από την, ε, το Ευρωκοινοβούλιο στη Γενική Διεύθυνση για την Περιφερική Πολιτική ακριβώς από την Επιτροπή Ρέτζι 2009 δόθηκε η εντολή. Η ιδέα ποια ήταν να υποστηριχθούν καινοτόμε και ολοκληρωμένες δράσεις ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πολυδιάστατο αυτό πρόβλημα το οποίο αναφύεται όσον αφορά την ένταξη των κοινοτήτων Ρωμά, των συγκάνων στις κοινωνίες μας διάφορες δραστηριότητες εντοπίστηκαν και ε, καθορίστηκε και ο προϋπολογισμός για αυτό το εγχείρημα 5 εκατομμύρια ευρώ ε, υποβάλαμε προσφο... Ε, άνοιξε η δυνατότητα υποβολής προσφορών είχαμε λοιπόν αρκετούς άξονες πάνω στους οποίους αναπτύξαμε αυτές τις δραστηριότητές μας ένας άξονας αφορούσε την πρώιμη παιδική ηλικία και περίθαλψη μετά ο επόμενος άξονας ε, η αυτοαπασχόληση με μικροδάνεια. Τρίτος άξονας ε, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση και ταυτόχρονα είχαμε άμεσες επαφές ε, με την παρακολούθηση και αξιολόγηση με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη 2010 και άλλες δραστηριότητες που σχετιζόντουσαν με τη συλλογή στοιχείων πάλι το 2010. Με άλλα λόγια προσπαθούσαμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προσπαθώντας να εξετάσουμε, να διερευνήσουμε αυτό το πεδίο σε αυτή την ε, δράση ώστε να υπάρχει πρόσθετη αξία που θα πέρε από αυτές τις δράσεις για το μέλλον. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι ότι θα τα εξετάσω ένα προς ένα αυτά τα κλονάρια, ας το αποκαλέσω έτσι, αυτής της δράσης μας. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο κλάδι, ο πρώτος κλάδος, πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την προεσπελασιμότητα για τα παιδιά των Ρωμάτων Τσιγκάνων, σε αναβαθμισμένες ε, υπηρεσίες στοχοθετημένη ομάδα παιδιά μέχρι 6 ετών ηλικίας, ηλικιακά. Η ιδέα που είχαμε ποια ήταν. Ήταν να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση των παιδιών αυτών, αυτής της ομάδα στόχου, στην ε, εκπαίδευση, σχολική εκπαίδευση αρκετά νωρίς, ε, πρώιμη πρόσβαση, ώστε να προετοιμάσουμε, να προελιάνουμε το έδαφος για αυτή την ε, σχολική παιδεία, εκπαίδευση και να προετοιμαστούν και οι μελλοντικέ προοπτικές. Πρώτα απ' όλα οι εταίροι. Ο κυριότερος εταίρος ήταν το Ταμείο για την εκπαίδευση των Ρωμά, των Τσιγκάνων είχαμε ε, εταίρους στο διεθνές και στο τοπικό επίπεδο. Συνολικός προϋπολογισμός περίπου 2 εκατομμύρια, γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ συνεισφορά Ευρωπαϊκής Ένωσης 1,9 ε, εκατομμύρια ευρώ. Οι εταίροι ήταν Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρωμανία και η πρώην ε, Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της ε, Μακεδονίας με 16 τοποθεσίες που είχαν επιλεγεί διάρκεια σχεδίου 24 μήνες, δύο έτη. 4.000 παιδιά μπόρεσαν να καλυφθούν από αυτό το πρόγραμμα με ηλικιακά μέχρι 6 ετών. Επίσης καταφέραμε να θεσπίσουμε καλές επαφές με αρκετούς μη κυβερνητικού οργανισμούς, ΜΚΟ, να έχουμε αηφόρου χαρακτήρα εταιρικέ σχέσεις όσον αφορά τα παιδιά των Ρώμα, των Τσιγκάνων σε αυτές τις δράσεις μας. Τούτων λεχθέντων κάποια από τα πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτού του τμήματος, ε, αυτού του σχεδίου, βλέπετε ότι ο στόχος ήταν να ε, αναβαθμιστεί η πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου ε, τέτοιες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Σε κάποιες χώρες καταφέραμε το 100% αυτού του περίγυρου. Ειδικά στη Σλοβακία καταφέραμε αυτό που προανέφερα ήταν Ουγγαρία, Ρουμανία 100%. Στη Σλοβακία για τις προσχολικές ε, δυνατότητες που θέλαμε να βελτιωθούν αποδείχθηκε ότι ήταν ε, μικρότερο το ποσοστό από τις ανάγκες όμως καταφέραμε το πλήρες δυναμικό που είχαμε να το αναπτύξουμε στην Φάιρομ, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με άλλα λόγια καταφέραμε αν όχι πλήρη συμμετοχή τουλάχιστον μερική συμμετοχή ώστε όλα αυτά τα παιδιά να μπορούσαν σε αυτές τις περιοχές στις οποίες δράσαμε να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ποια ήταν τα στοιχεία αυτά. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τη δυνατότητα να δράσουν ανεξάρτητα και να αυτενεργήσουν οι οικογένειες, κυρίως οι γυναίκες. Επίσης οι γυναίκες όσον αφορά την παρακολούθηση και συνοδευτικές δραστηριότητες, διότι αντιληφθήκαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στοχεύουμε στις ιδιαίτερες ε, ιδιομορφίες και χαρακτηριστικά της κάθε κοινότητας. Να δίνεται η δυνατότητα στις ίδιες τις κοινότητες των τσιγκάνων να συνοδεύουν και να, ε, συμπληρώνουν αυτές τις δραστηριότητες ασχοληθήκαμε και με την κατάτηση και εκπαίδευση ε, δασκάλων. Με μια πολιτική χωρίς αρνητικές ε, διακρίσεις. Μια ολοκληρωμένη ε, πολιτική ένταξης των ατόμων σε αυτήν για τη βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και με προσφέροντας επίσης και απογευματινά μαθήματα ή ε, προγράμματα. Προσπαθήσαμε να είμαστε το δυνατόν πιο καινοτόμοι δοκιμάζοντας ε, διάφορες δραστηριότητες. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία ήταν ε, η συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Τώρα, υπό τους όρους συμπερασμάτων αυτής της δράσης ξεχωριστά από το πιλωτικό αυτό σχέδιο το θετικό ήταν ότι καταφέραμε 100% για τις προσχολικές δραστηριότητες των παιδιών Ρωμά, των μικρών τσιγκάνων, να τις καλύψουμε. Καταφέραμε να διευρύνουμε και να επεκτείνουμε το δυναμικό, π.χ. στη Σλοβακία. Επίσης εισαγάγαμε κάποιες εναλλακτικές δραστηριότητες που ξεκίνησαν κάποιες από αυτές στη Σλοβακία αλλά και στη Ρουμανία καταφέραμε να, υπάρξουν, ε, να υπάρξει συνοδευτική δραστηριότητα όσον αφορά οικογένειες τσιγκάνων και να βελτιώσουμε το συσχετισμό μεταξύ των προσχολικών αυτών δυνατοτήτων και ευκαιριών και των οικογενειών τσιγκάνων. Υπάρχει ακόμα ευρύ περιθώριο, θεωρούμε, μεγάλο δυναμικό για βελτίωση στη συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Είναι μια βήμα προς βήμα σταδιακής ανάπτυξης ε, ε, εξέλιξη. Δεν μπορεί 100% διαμιάς να ε, επιτευχθεί. Πρέπει λοιπόν κλιμακούμενα βήμα προς βήμα να ε, ενταθεί και να αυξηθεί η δράση και η αποτελεσματικότητα. Επίσης η κινητικότητα να διευκολυνθεί. Με την επιτυχία αυτή του, πολι... του πιλωτικού προγράμματος θα πρέπει να τύχει συνέχεια ώστε να υπάρξει αηφορία ως προς τις ε, επιπτώσεις, τα αποτελέσματα. Ο επόμενος άξονας ήταν η αυτοαπασχόληση μέσω μικροδανείων. Ο προϋπολογισμός 1,6 ε, εκατομμύρια με ευρωπαϊκή συμμετοχή 1,4 εκατομμύρια. Οι οργανώσει των εταίρων από πλευρά οργανωτικής τι είχαμε είχαμε και τη συμμετοχή του Υπουργείου ε, Ανθρώπινων Πόρων της Ουγγαρίας. Ο στόχος ήταν να υποστηριχθούν οι κοινότητες των Ρωμάτων συγκάνων, να αυτενεργήσουν, να αυτοτελώς να ενεργήσουν, να ιδρύσουν μικροεπιχειρήσεις με μικροδάνεια. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στόχευε στην ε, ενδυνάμωση του δυναμικού μέσω, μικρο, μέσω μικροδάνεια και οι δύο αυτοί άξονες ξεκίνησαν τις δραστηριότητες τους το 2010. Ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες τους το 2012. Γι' αυτό μπορούμε να σας παράσχουμε τώρα πλήρη συμπεράσματα επ' αυτών των δράσεων. Παρότι πρέπει περαιτέρω να αξιολογηθούν ακόμα πιο εξειδικευμένα οι δράσεις αυτές. Τώρα, σε σχέση με τα δάνεια, για την, ε, να, ξεκινήσουν μικροεπιχειρήσεις στις ε, ε κοινότητες των συγκάνων. Αυτό θα είναι αρκετό για να υπάρξει εισόδημα το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί αυτά τα δάνεια αλλά και θα παράγει πρόσθετο εισόδημα για τις ανάγκες των οικογενειών αυτών των συγκάνων. Συμπεράσματα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό ως, πολι... ως πιλωτική δράση. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι για κάποιες από αυτές τις δράσεις πρέπει διαφορετική προσέγγιση να ακολουθηθεί. Κάποιες προσεγγίσεις ε, υιοθετήθηκαν ε, που αλλού, ε, όχι σε κοινότητες τσιγκάνων εφαρμόστηκαν, φάνηκε και αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επαρκή αυτά και ότι για παράδειγμα με μια ομάδα στόχου ξεκινήσαμε στην αρχή και στο μεσοδιάστημα έπρεπε να αλλάξει η στοχομάδα διότι αντιληφθήκαμε ότι για να μπορέσουμε να έχουμε μια ελάχιστη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις δράσεις μας έπρεπε να στοχοθετήσουμε εκείνους τους Ρωμά, τους, πιο, τους που δεν ήταν οι πιο φτωχοί αλλά που είχαν κάποια ε, επιχειρηματική δράση στο παρελθόν έπρεπε να συνδυαστούν αυτά με δυνατότητες ε, επιμόρφωσης Κατάρτιση, κατάρτισης, εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν πιο εξειδικευμένα να καταρτιστούν προηγούμενα αυτά τα άτομα για την επιχείρηση που θα ξεκινούσαν. Να αποκτήσουν χρηματοοικονομικές γνώσεις, ώστε η επιχείρηση που θα άνοιγαν να, μπορέσει, να μπορούσε να στεφθεί με επιτυχία. Επίσης, ε, εξετάσαμε τις δυνατότητες ε, και σε σχέση και με ε, την κατάρτιση επιτόπου των ατόμων αυτών. Όμως όλα αυτά κατέστησαν δαπανηρά αυτό το εγχείρημα. Στο τέλος τέλος βλέποντας ποιο ήταν το input και ποιο ήταν το output πραγματικά φαίνεται ότι ήταν ίσως κάπως πολύ δαπανηρό αυτό το εγχείρημα και ίσως τόσο, όχι τόσο αποτελεσματικό σε σχέση με τα κονδύλια που διατέθηκαν. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο θα έλεγα ε, θετικά. Σε σχέση λοιπόν με αυτά τα οποία έγιναν πρέπει ε, μπορούμε να ε, γνωρίζουμε πλέον ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να συνδυάζονται με άλλες παράλληλες δραστηριότητες για να είμαστε πιο επιτυχείς βλέπει κανείς έτσι στη συνέχεια τα αδύναμα στοιχεία τα οποία εντοπίστηκαν, τα πιο ευάλωτα σημεία, σε σχέση για παράδειγμα και με τη συνεργασία με τις τοπικές ή εθνικές αρχές. Κέρια σημασία σε αυτό το σημείο και φάνηκε σε αυτό το συγκεκριμένο πιλωτικό σχέδιο το οποίο ξεκινήσαμε ότι δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί στη διαμόρφωση αυτών των σχέσεων. Αν έχετε κάποια ερώτηση για κάποιο από αυτούς τους συγκεκριμένους άξονες, είμαστε πρόθυμοι να ε, δώσουμε απαντήσεις. 400 ετούντες ε, ήταν εκείνοι που προσπαθήσαμε να καλύψουμε αλλά 338 ήταν εκείνοι που καταφέραμε να καλυφθούν στο τέλος σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του έργου μας. Ο επόμενος άξονας ε, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση ενημέρωση, πληροφόρηση ευαισθητοποίηση. Ο τίτλος ήταν «React», ε, αντιδράστε, να κάνουμε την Ευρώπη έναν χώρο που θα είναι ε, δίκαιος για τους Ρωμά, τους Τσιγκάνους. Συνολικός προϋπολογισμός 1 εκατομμύριο ευρώ. ευρώ. Στόχος ήταν να αλλάξουν οι αρνητικές ε, τοποθετήσεις και οι προκατηλημένες απόψεις εναντί των Τσιγκάνων και να υπάρξει ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα των Τσιγκάνων ε, συνεισφέροντας πως οι χώρες σε οποίες εμπλακή, ε, υπήρξε εμπλοκή ήταν η Ρουμανία, η Ιταλία, Βουλγαρία και Αλβανία αμέσως φυσικά ε, συνειδητοποιήσαμε ότι τέτοιου είδους εκστρατείες ε, δεν μπορούν να ε, είναι αυθύπαρκτες. Πρέπει να συνδυάζονται και με μια παρουσίαση, μια αποτελεσματική παρουσίαση των επιτευγμάτων και των δράσεων για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Κάποια από τα συμπεράσματα από αυτή την πρωτοβουλία που αναπτύξαμε θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής. Είχαμε κάποιες εκστρατείες ε, και σε σχέση και με ε, επιτόπου δράσεις. Προσπαθήσαμε να βρεθούμε στο επίκεντρο της προσοχής ε, των πολιτών. Είχαμε και προσωπικότητες, εξέχουσες προσωπικότητες που εμπλέξαμε συνεργαζόμενοι με αυτές τις προσωπικότητες για αυτές τις εκστρατείες. Είχαμε και βιντεοκλίπ, κινητοποιήσαμε και τα κοινωνικά media, social media, είχαμε και επιτόπου την καλύτερη ας το ε, εμπλοκή ομάδων advocacy groups για την προβολή αυτών των ε, ε, δραστηριοτήτων είχαμε συνολικά στην ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων μας θετικά αποτελέσματα. Επιτόπου συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους και ενώσεις ε, επίσης ε, φυσικά ταυτοποιήσαμε, εντοπίσαμε ότι για να υπάρχει αηφορία και να υπάρξει αποτελεσματική μάζα δράσης θα πρέπει πιο μακροπρόθεσμα να διεξάγονται τέτοιου είδους ε, δράσεις και θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό ιστό. Από κοινού λοιπόν με τις ΜΚΟ, τις ΜΚΟ για τους Ρωμά, για τους Τσιγκάνους πρέπει να εντάσσονται και αυτές στις δράσεις μας εξίσου όπως ε, και από πλευράς μας έτσι και από πλευράς τους αμφίδρομα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό μπορεί να συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση και κατά, των ρατσιστικών τάσεων π.χ. επιτόπου στη Ρουμανία. Στο τέλος εν κατακλείδη θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι. Κάποιες συνολικότερες ε, πολιτικές μαθήματα που μπορέσαμε να συναγάγουμε συνολικότερα από αυτό το εγχείρημα. Ένα από τα θετικά αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος που πραγματικά μέσα από όλη αυτή τη δράση επετεύθη για τη διεύρυνση της, ε, του καλύτερου συντονισμού, των μηχανισμών συντονισμού των αρμόδιων για τα θέματα των συγκάνων, αυτό είναι κάτι σημαντικό και για σήμερα κιόλα έχουμε συναδέφους παρόντες από τις διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, αποτελούν ανάγλυφα απόδειξη αυτής της ε, κοινή προσπάθειας συντονισμού. Πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπορούν στο ευρύτερο ε, εύρος να συμμετάσχουν σε αυτές τις δράσεις, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού, των, τους μεγαλύτερους πληθυσμούς τσιγκάνων. Επίσης εντοπίσαμε, ταυτοποιήσαμε τα συμπεράσματα και μαθήματα εκείνα που θα θέλαμε να εισαχθούν την περαιτέρω μετεξέλιξη αυτών των προγραμμάτων μετά το 2014 σε ένα χρονορίζοντα. Μαθήματα που συνδέονται και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και σχετικές δράσεις, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης και των σχετικών δράσεων που προβλέπονται από τα κονδύλια του. Η γνώση που καταφέραμε να αποκομίσουμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει πραγματικά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Συντοπίσαμε δηλαδή ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά στοιχεία και καταφέραμε επίσης να θεσπίσουμε μία βάση για τις μελλοντικές μας δραστηριότητες. Μέσω του πιλωτικού λοιπόν αυτού και παράλληλα με το πρόγραμμα αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε αρκετές γνώσεις προκειμένου να καταφέρουμε να τροποποιήσουμε το εφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα διορθωτικά ταμεία για την περίοδο 2007-2013. Και επίσης καταφέραμε να εισαγάγουμε την επωνομαζόμενη δραστηριότητα Integrated Housing στέγαση για την συμπερίληψη, την ένταξη των Ρωμά. Μέσω της συλλογή των δεδομένων και μέσω της επεξεργασίας τους καταφέραμε να συλλέξουμε πάρα πολλά δεδομένα. Επίσης γίνανε πολλές έρευνες. Καταφέραμε λοιπόν μέσω των ενεργειών αυτών και μέσω της συγκέντρωσης κυρίως δεδομένων να δημιουργήσουμε μια πάρα πολύ καλή βάση για τις μελλοντικέ μας δραστηριότητες και καταφέραμε επίση να πτύξουμε και διάφορες μεθόδους προκειμένου να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας για την υποστήριξη των κοινοτήτων Ρωμά. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών καταφέραμε να συνεργαστούμε πολύ αποτελεσματικά με το Πρόγραμμα Ανάπτυξη των Εθνών, με την Παγκόσμια Τράπεζα, με την Υπηρεσία των Οργανισμών για τη Θεμελιώδη Δικαιώματα και μια πολύ σημαντική έρευνα δημοσιεύτηκε για την ε, κοινωνική-οικονομική κατάσταση των Ρωμά τον Απρίλιο Μία τελευταία διαφάνεια που έχει να κάνει πάλι με τα διδάγματα τα οποία αντλήσαμε μέσω του προγράμματος αυτού. Είδαμε εδώ πέρα ότι πραγματικά μπορεί να υπάρχει μία διασύνδεση ανάμεσα στο πρόγραμμα αυτό και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Ρωμά. Ουσιαστικά θέλουμε να δημιουργήσουμε εδώ πέρα τις βέλτιστες δυνατές συνέργειες ανάμεσα στις δράσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό στη νέα γενιά προγραμμάτων να χρησιμοποιήσουμε τη διασύνδεση αυτή, τις συνέργειες αυτές και να συνδεθούν και με τα ταμεία επενδύσεων, τα επενδυτικά ταμεία. Ξέρετε ότι στη νέα περίοδο προγραμματισμού μια βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει μια σωστή εθνική στρατηγική για την ένταξη των δρομάτων σε επίπεδο κράτους μέλους λοιπόν. Πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε όμως να αυξήσουμε την κλίμακα αυτή των βέλτιστων πρακτικών, των καλών αυτών δαγμάτων που έχουμε αντλήσει, πώς θα καταφέρουμε να τα εντάξουμε στη νέα περίοδο προγραμματισμού και να εναρμονίσουμε τις πρακτικές αυτές για όλα τα κράτη-μέλη. Προκειμένου λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο, στις 15 ε, Μαρτίου του 2013 θα διοργανηθεί μια συνδιάσκεψη, βασικός στόχος της οποίας είναι να ε, διαβιβαστούν, να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αποτελέσματα, τα πορίσματα αυτού του πιλωτικού προγράμματος και να καταφέρουμε να φέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο μαζί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που θα καταφέρουν να συζητήσουν κατά αυτόν τον τρόπο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θεωρώ ότι από άποψη θέσπισης πολιτικής το πρόγραμμα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί μάθαμε πολλά σημαντικά πράγματα και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σας πω ότι είναι διαθέσιμα και τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι παρόντα εδώ για να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε ο κύριος Τσέλερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, έκθεση αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ επίσης και για το πιλωτικό πρόγραμμα. Είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν εύκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Ξέρετε ότι τα πιλωτικά προγράμματα έχουν ως στόχο να αυξηθεί το επίπεδο γνώσης. Η γνώση βέβαια που κερδίσαμε εδώ πέρα δεν είναι νέα, απλώς επιβεβαιώθηκαν κάποια πράγματα με τρόπο εντυπωσιακό. οι κοινότητες των Ρωμά θα βρεθούν σε καλύτερη θέση αν όλη η κοινωνία τελικά των χωρών στις οποίες ζουν οι Ρωμά πραγματικά συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα και αν πραγματικά υποστηρίξουν όλοι τα προγράμματα αυτά. Και το είπατε και οι ίδιοι ότι ένα από τα δύναμα σημεία, τουλάχιστον σε μία χώρα στην οποία αναφερθήκατε, ήταν ότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα για αποτελεσματική συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Ε, άμα δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση δεν μπορεί να λυθεί κανένα πρόβλημα. Πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε στις κοινότητες των Ρωμά εταίρους, συνομιλητές, άνθρωποι που θέλουν να προωθήσουν τα προγράμματα ένταξης των Ρωμά. Ξέρετε ότι ε, στην δική μου την πόλη, στο Βερολίνο, έχουμε χιλιάδες Ρωμά. Άνθρωποι οι οποίοι ε, φύγαν από τις χώρες τους ακριβώς επειδή διώκονταν εκεί πέρα. Ήταν θύματα διακριτικής μεταχείρισης. Έρχονται όμως ως ε, Ρουμάνοι, Ούγγροι πολίτες στο Βερολίνο. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να συνεργαστούμε καλύτερα μαζί τους. Μέχρι στιγμής δυστυχώς η συνεργασία είναι πολύ περιορισμένη. Τα προβλήματα εκκρεμούν, υφίστανται ακόμα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φτάνουν στο Βερολίνο, αλλά δεν είναι καταλήλως προετοιμασμένοι. Έρχονται στο Βερολίνο και ουσιαστικά προσπαθούν να επιβιώσουν. Ζούνε σε κάποια τμήματα της πόλης τα οποία είναι αρκετά υποβαθμισμένα, πλήττονται από φτώχεια. Και μολονότι υπάρχουν κάποια κονδύλια και μολονότι προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, δεν το καταφέρνουμε πάντα. Βλέπουμε ότι πολλές φορές σε κάποια διαμερίσματα μικρά, σε διάρκεια, ζουν 60 άτομα μαζί. Υπό αυτές τις συνθήκες καταλαβαίνετε ότι τα πάντα γίνονται προβληματικά. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο, οι γονείς δεν νοιάζονται για την εκπαίδευση των παιδιών και το καθεξής. Το πρόβλημα λοιπόν των Ρωμά δεν έχει να κάνει μόνο με τις χώρες προελευσής τους, αλλά αφορά όλη την Ευρώπη. Συλλογικά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα των Ρωμά δίνοντας τα απαραίτητα χρήματα. Το σύνολο λοιπόν της κοινωνίας, τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στις υπόλοιπες χώρες, πρέπει να κινητοποιηθεί προκειμένου να καταλήξουμε σε μια νέα προσέγγιση για την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, για την κατάλληλη ενημέρωση των πολιτών και όπως σας είπα πρέπει να βρούμε και κάποιους συνομιλητές από την ίδια την κοινότητα των Ρωμά, κάποιους εκπροσώπους των Ρωμά, οι οποίοι να θέλουν και αυτοί να επιφέρουν κάποιες αλλαγές στην κατάστασή τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Αλφονσί. Ε, καταρχάς, πρέπει να εκφράσω την ικανοποίησή μας ε, και για το ότι ξεκίνησε αυτό το πιλωτικό σχέδιο από την Επιτροπή και γιατί το υλοποίησε η Επιτροπή σε μια σύντομη χρονική περίοδο. Νομίζω ότι ο απολογισμό είναι εύγλωτος. Η προσέγγιση είναι ενδιαφέρουσα και είναι σήμερα αναγκαίο να ξεκινήσουμε από αυτά που επιτεύχθηκαν για να προχωρήσουμε περαιτέρω και να αγγίξουμε κοινότητες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, τροτές, γιατί βρίσκονται σε μια κατάσταση πλήρους ε, τροτότητας. Και διότι οι κοινότητε στον Ρώμα θα πρέπει να μπορέσουν να έχουν μια ποιότητα ζωής όπως αυτή όλων ε, των υπολείπων πολιτών της Ένωση. Η Επιτροπή μας μπορεί νομίζω να παίξει ένα μικρό ρόλο πήγαινοντα λίγο παραπέρα. Λίγοι είμαστε εδώ σήμερα, κρίμα. Θα ήταν ε, ενδιαφέρον τα θέματα να αντιμετωπιστούν καλύτερα, ίσως με μια ακρόαση των εμπλεκομένων, ίσως με μια συνάντηση με μικιό με εκπροσώπους της κοινότητας των Ρωμά, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο πρόγραμμα αυτό, γιατί πιστεύω ότι η ανάδειξη και επικοινωνία των αποτελεσμάτων είναι κομμάτι της αποτελεσματικότητάς μας. Ο κύριος Βανίστελ ε, Ευχαριστώ. Πάντα θέμα επιλογών είναι όταν οι πολιτικές ομάδες ε, ξεκινούν με πιλωτικά σχέδια προσπαθώντας να δώσουμε έμφαση στις διαστάσεις εκείνες που συνδέονται με την περιφερειακή πολιτική και παρέχουν τη δυνατότητα να φτάσουμε σε υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων. Είδαμε σε πολλές περιπτώσεις επισκέψεων σε περιοχές με Ρωμά ότι θα έπρεπε να έχουμε μία πιο εστιασμένη προσέγγιση με μία πιο μακροχρόνια υποστήριξη. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει ενοποιημένη προσέγγιση, δεν θα λειτουργήσει. Ποιο είναι το θέμα. Είπαμε ότι οι κανονισμοί για... άλλαξαν το 2010 για τις ευάλωτες ομάδες με ιδιαίτερο στόχο τους Ρωμά. Τώρα, το έργο αυτό είναι προστιθεμένη αξία, αλλά υπάρχει. Πώς προχωράει το mainstreaming. Αυτό που δεν έγινε είναι τα κονδύλια που θέτουμε μέσω του Περιφερειακού Ταμείου, του Κοινωνικού Ταμείου, δεν αντλήθηκαν για τους Ρωμά. Ήταν τόσο δύσκολο να γίνουν, ε, να υπάρξει αποδοχή για να μπει αυτή η ομάδα ενοποιημένα ως προτεραιότητα, ούτως ώστε οι δυνατότητες και οι δράσεις αποκλίνουν πάρα πολύ. Δείτε τη Ρουμανία. Υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό άντληση περιφερειακών ταμείων, περιφερειακών πόρων. Ενώ είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πρόβλημα στους πληθυσμούς Ρωμά. Μπορεί να μας πει η Κομισιόν πώς μπορεί να παραταθεί το πρόγραμμα αυτό τα επόμενα χρόνια ή πώς μπορεί να γίνει καλύτερα το mainstreaming. Μαθαίνω κι εγώ αυτή τη στιγμή και προσπαθώ Προσπάθησα να κατεβάσω αυτή την εικόνα που έχετε στην ιστοσελίδα μου, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση πρέπει να γίνει πολύ μικρή. Πώς νομίζετε ότι άμα είναι τρεις γραμμές η ηλεκτρονική σελίδα θα ε, μπορέσει κάποιος να την αντιγράψει. Βάλτε τη διεύθυνση ε, ε, στο φυλάδιο. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ πέρα. Η επικοινωνία είναι σημαντική. Το δουλεύει η κυρία Κρούς, αλλά όλοι στην Επιτροπή θα πρέπει να έχουν υπόψη τους την επικοινωνία. Αυτό είναι μισό πράγμα. Δεν είναι πιστικό. Ξέρεις, για να τα κάνεις αυτά πρέπει να είσαι 16χρονος. Ε, καλύτερα να απαντήσετε στο τέλος, Επιτροπή. Ο Βλαντιμίρ Μάνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξαιρετικές οι δραστηριότητε αυτές. Συγχαρητήρια για τα πιλωτικά αυτά σχέδια, τα οποία συχνά παρέχουν την καλύτερη εμπειρία για μας. Είναι μια καλή αφετηρία για το μέλλον. Ίσως να είναι προβληματικό το να εξασφαλίσουμε ότι τα έργα αυτά παραμένουν βιώσιμα. Σε ό,τι με αφορά, δεν ξέρω να υπάρχουν πραγματικά βιώσιμα εγχειρήματα στον τομέα αυτό. Εγώ δουλεύω αρκετά με την κοινότητα αυτά και είναι σημαντικά να δώσουμε έμφαση στα παιδιά. Να στηρίξουμε τα παιδιά καθοδόν μέχρι να βρουν δουλειά. Χρειαζόμαστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά Ρωμά για να μπορέσει να είναι βιώσιμη μια λύση με απέναντι, τους. Χρειάζεται να δουλέψουμε με, την τοπή, με τους Δήμους. Και συμφωνώ ότι οι Δήμοι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί από ότι οι κυβερνήσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν δήμαρχος μιας πόλης, με είχε προσεγγίσει ένας ε, Ρωμά που μου ζήτησε τη βοήθεια για να βρει δουλειά. Το ρώτησε τι μπορείς να κάνεις και μου είπε έχω αποφυτίσει από ε, ένα οδείο, παίζω βιολί. Τον έστειλα σε μία εκδήλωση που οργάνωνε η πόλη μας, έπαιξε εξαιρετικά και τώρα είναι ε, διευθυντής μιας μικρής ορχήστρας. Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν είναι να δώσουμε υποστήριξη και να παράσχουμε εκπαίδευση, να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο από τον νωρί μέχρι τέλος και να τους συνοδεύουμε, να τους παρακολουθούμε, να τους προσφέρουμε θέσεις εργασίας με έναν βιώσιμο τρόπο. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζονται δύο γενιές Ρωμά για να γίνει κάτι τέτοιο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα αναφερθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο και συγχαίρω επίσης φυσικά τον κύριο Τσέρερ για τις απόψεις που εξέθεσε και τους άλλους συναδέλφους. Πολύ συχνά μιλάμε για το πρόβλημα των συγκάνων, των Ρωμά, ως πρόβλημα των χωρών προέλευσης. Μετά το, ως πρόβλημα των χωρών υποδοχής. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να ομιλούμε για το θέμα των συγκάνων ως ευρωπαϊκό ζήτημα. Είναι η μόνη προσέγγιση, αν υιοθετήσουμε αυτήν, που θα δώσει αποτελέσματα. Ευρωπαϊκό ζήτημα λοιπόν η Τσιγκάνη. Δεύτερη παρατήρηση και είναι πολύ σημαντικό και αυτό αξιότιμοι συνάδελφοι. Το θέμα της επόμενης γενιάς Τσιγκάνων των Ρωμά να ε, επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό. Η Ρωμά, η Τσιγκάνη στη Ρουμανία, στη χώρα μου για παράδειγμα που για παράδειγμα το 1990 κατά την αλλαγή του καθεστώς, καθεστώτος ε, που ήταν 17 ετών κατά την αλλαγή στη Ρουμανία σήμερα είναι 23 ετών και αυτό τι και άλλοι Ρωμά έχουν ολοκληρώσει τις ε, σπουδές τους ε, σε πανεπιστήμια. Είναι η προσωπική μας αυτή η εμπειρία όσον αφορά τη Ρουμανία αλλά και σε άλλες ε, χώρες προέλευσης μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτό. Αυτή η νέα λοιπόν γενιά των τσιγκάνων που έχουν ήδη αποφοιτήσει από πανεπιστήμια, αυτή η νέα γενιά είναι η κινητήρια δύναμη για να αλλάξουν τα πράγματα σε σχέση με τους τσιγκάνους. Φυσικά αρκετοί από αυτούς επιλέγουν να μην ταυτοποιούνται πλέον με την κοινότητά τους ως τσιγκάνοι και την εγκαταλείπουν, φεύγουν, αποχωρούν από αυτήν, όμως θα μπορούσαν ε, τέτοιου είδους άνθρωποι να είναι οι κινητήρες για την αλλαγή νοοτροπίας και την αλλαγή ε, της κατάστασης και προσέγγισης των τσιγκάνων. Τώρα, δεν θέλω να εμείνω και να περι, ε, περισσότερο σε σημεία που έχουν καλυφθεί από τους άλλους συναδέλφους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι θα πρέπει να μιλήσουμε μιλήσουμε για αυτές τις δράσεις. Πιλωτικά σχέδια για παράδειγμα, όπως αυτά για τα οποία ακούσαμε, πρέπει να αξιολογηθούν και να δούμε τις δυνατότητες να υπάρξουν μόνιμες χρηματοδοτήσεις και μόνιμα διαρκέστερα προγράμματα και να γνωρίζουμε αυτή την προοπτική να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι κάνουμε λόγο για ολόκληρες δεκαετίες. Δεν ξέρω, είμαι μηχανικός, μηχανολόγος. Δεν πρέπει να αναφερόμαστε μόνο σε κάποιες δεκαετίες, να δούμε πιο μακροπρόθεσμα πώς θα δώσουμε συνέχεια. Τότε θα στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα, αν είναι πιο μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Μωρίς Πόγκα, παρακαλώ. Euh, Όχι, δεν θέλετε να παρέμβετε. so that's, that's εσείς είσαστε λοιπόν αυτοί που παρενέβησαν και εγώ να προσθέσω μια ερώτηση για τη συλλογή δεδομένων που κάνατε με το δικό σας όργανο και άλλα όργανα. Αυτό το δημοσίευμα ή αυτή η επισκόπηση ότι οποιοδήποτε και αν ήταν αυτό το δημοσίευμα την προηγούμενη τελευταία άνοιξη που δημοσιεύθηκε ήταν μια ξεχωριστή δραστηριότητα εξάπαντος ή ξεκινά και μια νέα ή συνεχίζεται άλλη δραστηριότητα για αυτή την συλλογή δεδομένων. Δεύτερη ερώτηση, μια πρόταση από τον Φρανσουά Αλφονσί να υπάρξει μια ευρύτερη ακρόαση που θα διεξαγόταν εδώ στο, στους κόλπους της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής με πρόσκληση που θα απευθυνόταν και θα προσκαλούσαμε και άλλα θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, και ιδιαίτερα εκείνε που ασχολούνται περισσότερο με του τσιγκάνου και οι εκπροσώπου τη ίδια τη κοινότητα των τσιγκάνων. Ε, ε, το εξετάζουμε αυτό. Εσεί όμω από πλευρά Επιτροπή έχετε συντονισμό των δραστηριοτήτων σε σχέση με την ε, Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, Γενική Διεύθυνση για τι Περιφέρειε, μέσα από το συντονιστικό αυτό έργο υπάρχει κάποια άλλη τέτοια προοπτική. Υπάρχουν πολλέ άλλε δραστηριότητε νομίζω νομίζω. Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε σε μια τέτοια ακρόαση φυσικά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερώτησή μου, αυτά τα συμπεράσματα, αυτά τα μαθήματα τα οποία συνάγονται από αυτό το ε, πιλωτικό πρόγραμμα. Μίλησε ο Λαμπέ Φανίστερ Ρο για την ένταξη όλων αυτών των προοπτικών στις ευρύτερες πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ το βλέπετε εσεί αυτό. Θα μπορούσε να ενταχθεί μέσα στις ε, κανονικές δραστηριότητες ε, όσον αφορά την, ε, τα θέματα περιφερειών ή προβλέπετε γίνεται ανάληψη κάποιας καινοτόμας δράσης από πλευράς ε, της Γενικής Διεύθυνσης ε, για την ε, Περιφερειακή Ανάπτυξη και τις Περιφέρειες. Κάτι που θα συντόνιζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρξει συνοδευτική δραστηριότητα σε σχέση με αυτό το πιλωτικό σχέδιο ή θα ενταχθούν μόνο τα συμπεράσματα μέσω κανονισμών και δράσεων στο επίπεδο κρατών μελών και περιφερειών και πόλεων. Πώς το βλέπετε αυτό. Ευχαριστώ. Και μπορούμε και τις διαφάνειες να τις έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή και εμείς επιπρόσθετα σε σχέση με τον Λάμπερτ που τα έχει ήδη στη διάθεσή του, θα θέλαμε και την ηλεκτρονική τους μορφή να μας διαθέσετε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις παρατηρήσεις και τις πολύ καλές ερωτήσεις σας. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι ευρωβουλευτές είναι ικανοποιημένοι με το πιλωτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ουσιαστικά θεωρείται ότι ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δίγησε πολύ καλά συμπεράσματα και διδάγματα. Οι παρατηρήσεις ήταν πολύ καλές όσον αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά να μην αναφερόμαστε μόνο στα ζήτημα, σε ζητήματα της στέγασης, αλλά το ζήτημα αυτό να συνδέεται με την εκπαίδευση, με την ενδυνάμωση της ε, κοινότητας των Ρωμά προκειμένου να καταφέρουν να ξεκινήσουν μια επαγγελματική δραστηριότητα, να βρουν μια θέση εργασίας. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πιλωτικά προγράμματα τελικά επηρεάζουν πάρα πολύ και την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου όπου για παράδειγμα τα όσα προβλέπονται για τη στέγαση θα πρέπει να είναι πλέον προγράμματα ολοκληρωμένα, να μην αναφέρονται μόνο δηλαδή στη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, αλλά να συνδέεται η δημιουργία των κατοικιών αυτών και με άλλε δραστηριότητε. Και βέβαια θα πρέπει να προβλέπετε και χρηματοδότηση για όλα αυτά, όπω είπαμε. Είπατε επίση ότι δεν χρησιμοποιούνται πάρα πολλοί πόροι μέχρι στιγμή. Και πολλοί ευρωβουλευτέ μα ρώτησαν Πώ θα εξελιχθούν στο μέλλον οι δραστηριότητε αυτέ για του Ρωμά, θα ευθυγραμμιστούν κατά κάποιο τρόπο, θα εξορθολογιστούν. Κοιτάξτε, Όλα αυτά τα διδάγματα τα οποία έχουμε αντλήσει αποτελούν αυτή τη στιγμή αντικείμενο αξιολόγηση για να δούμε τελικά πώ θα καταφέρουμε να θεσπίσουμε και να εφαρμόσουμε μελλοντικά προγράμματα. Θέλουμε λοιπόν να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα διδάγματα, από την άλλη όμω είμαστε και Δεν μπορούμε τόσο εύκολα να πάμε από το πιλωτικό πρόγραμμα σε κάτι το οποίο θα ισχύει σε όλε τι χώρε. Θέλουμε προφανώ να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή του προγράμματο αυτού το είπατε κι εσείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια διασύνδεση με την ε, τοπική αυτοδιοίκηση, με τους ε, εκπροσώπους των Ρωμά και τους άλλους εμπλεκομένους σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Ήδη έχουμε ε, θεσπίσει κάποιες πολύ καλές πρακτικές, αλλά απομένουν ακόμα να γίνουν πολλά. Πρωτού τελικά ότι μπορούμε να πετύχουμε την ε, ένταξη των προγραμμάτων αυτών σε διάφορες πολιτικές. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τις καλές πρακτικές που έχουμε από το πιλωτικό πρόγραμμα και προσπαθούμε να δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να εντάξουμε τις πρακτικές αυτές στη νέα περίοδο προγραμματισμού. Ξέρουμε τώρα ποια είναι τα μοντέλα, ποια είναι τα πρότυπα τα οποία λειτουργήσαν καλά και ποια όχι. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αποφύγουμε. Ορισμένοι είπατε ότι θα θέλατε να δείτε εδώ πέρα και τους ίδιους τους δικαιούχους του προγράμματος αυτού προκειμένου να μας πούνε και οι ίδιοι από πρώτο χέρι ποια ήταν η εμπειρία τους. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι δικαιούχοι έχουν κάνει ήδη συστάσεις πολιτικής, περιλαμβάνονται στο πιλωτικό πρόγραμμα και δώσαμε πάρα πολύ προσοχή σε αυτό το τμήμα, να ακούσουμε δηλαδή και τους δικαιούχους. Θα πρέπει εσείς όμως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθείτε περισσότερο και όντως σας ενθαρρύνουμε να διοργανώσετε μια δημόσια ακρόαση και να καλέσετε όλους τους εμπλεκομένους και τους εκπροσώπους της κοινότητας των Ρωμά. Τώρα το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό δεν λειτουργήσε πάρα πολύ σε κάποιες χώρες. Αυτή τη στιγμή θεσπίστηκε το πρόγραμμα, έρθαμε σε επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση και έχουμε ξεκινήσει κάποιες δραστηριότητες και έχουμε ενώσει ουσιαστικά τις δυνάμεις μας με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την Παγκόσμια Τράπεζα με την ε, Τράπεζα Ανάπτυξη Συμβουλίου της Ευρώπης, με όλες τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες στις δραστηριότητές μας όσον αφορά τη δημιουργία ικανοτήτων, capacity building σε τοπικό επίπεδο, γιατί καταλάβαμε τελικά ότι αυτός είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία θα καταφέρουμε να εντάξουμε αυτή τη διάταξη των Ρωμά στι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση, αν καταφέρουμε τελικά να εμπλέξουμε περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, ποια θα είναι η προσέγγιση του ζητήματο αυτού στο μέλλον. Ήδη στα έγγραφα που έχουν παρουσιάσει οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπής, στα position papers, προτείνεται να ξεκινήσει ένα άτυπο διάλογο με τι εθνικέ αρχέ. Το ζήτημα λοιπόν αυτό ήδη υφίσταται, θεωρείται οριζόντιο ζήτημα και ήδη το βλέπουμε στην εξάντε αιρεσιμότητα. Έχει τεθεί δηλαδή ως προϋπόθεση σε διάφορα προγράμματα. Αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, με την αστική ανάπτυξη. Ξέρετε ότι πάρα πολλά ζητήματα των Ρωμά έχουν να κάνουν με υποβαθμισμένες φτωχές αστικές περιοχές. Προσπαθούμε λοιπόν τις σχετικές αστικές δραστηριότητες να τις εντάξουμε όλες σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Επίσης προσπαθήσαμε να κάνουμε μια χαρτογράφηση της φτώχειας. Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει και τα οποία συνδέονται με την ένδυα. Έχουμε διάφορα στατιστικά δεδομένα σε διάφορα επίπεδα, τα οποία όμως δεν καταφέρουν να καταδείξουν τα πραγματικά προβλήματα των, των Ρωμά. Γι' αυτό το λόγο κάναμε και αυτή την ε, χαρτογράφηση της ένδυας προκειμένου να δούμε ακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι θύλακες φτώχειας που υπάρχουν στις διάφορες περιοχές. Έτσι θα καταφέρουμε μόνο να βοηθήσουμε πραγματικά τους Ρωμά. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερη συνεργασία, συντονισμό προγραμμάτων για να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά προγράμματα του main, ε, αποτελέσματα με του mainstreaming στη νέα περίοδο προγραμματισμού. Τώρα, όσον αφορά την ιστοσελίδα που είπατε, θα μιλήσω με τους ανθρώπους που ασχολούνται με την υπηρεσία πληροφορικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διορθώσουν το πρόβλημα το οποίο θίξατε. Πάντως, θα σας συνιστούσα είτε εσείς ίδιοι προσωπικά, είτε μέσω εκπροσώπων σας να συμμετέχετε στην συνδιάσκεψη αυτή που θα διοργανώσουμε, γιατί πιστεύω ότι θα καταφέρετε πραγματικά να δείτε πώς ένα πιλωτικό πρόγραμμα μπορεί τελικά να εμπνεύσει επίσημα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να απάντησα σε όλους. Ναι, ξέχασα και μία ερώτηση Κυρία Πρόεδρε, εσεί αναφερθήκατε στι εκθέσει. Μα είπατε αν η έκθεση του Απριλίου ήταν η μοναδική όχι. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πάρα πολλέ εκθέσει του UNDP, τη Παγκόσμια Τράπεζα, που έχει μια έκθεση που έχει συνταχθεί με του δύο αυτού φορεί και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση του ευάλωτου χαρακτήρα των, κοινοτών, των κοινοτήτων Ρωμά και για την καλύτερη ένταξή του στην Ανατολική Ευρώπη, έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τον 2012 και μία άλλη η οποία αναφέρεται στο πώς μπορεί να κλείσει το χάσμα αναλφαβητισμού ή ε, μη συμμετοχή των πολύ μικρών παιδιών Ρωμά στα νηπιαγωγεία και τα σχολεία. Σε κάθε περίπτωση μέσω των μελετών αυτών προσπαθούμε να δούμε ποια κενά γνώσεις έχουμε, πού πρέπει να μάθουμε περισσότερα πράγματα προκειμένου να συμπληρώσουμε καλύτερα τα προγράμματα ένταξης των Ρωμά. Και ξέρετε ότι υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων για τους Ρωμά. Και ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσουμε όλα αυτά τα εθνικά προγράμματα, τα προγράμματα τα οποία θα υποβάλουν τα κράτη-μέλη και ελπίζουμε ότι μέσω των προγραμμάτων αυτών και εφόσον γίνει καλή επιλογή προγραμμάτων θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των Ρωμά. Δεν ξέρω αν κάποιο αδερφό μου θέλει να πάρει το λόγο. Να πω και κάτι ακόμα όσον αφορά την ε, μη καλή εφαρμογή των προγραμμάτων σε κάποιες χώρες. Αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι σε όλα τα κράτη-μέλη που είναι χώρες προέλευσης για τους Ρωμά, προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με τις τοπικές αρχές προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε καλύτερα τα προγράμματα τα οποία έχουν για τους Ρωμά. Πρόεδρος, οι συνάδελφοι από τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουν να πάρουν το λόγο. Αν όχι, τότε έχω μια παρατήρηση ακόμα να κάνω. Διαπραγματευόμαστε τώρα τους μελλοντικού καονισμούς και τίθεται το ζήτημα των συμφωνιών εταιρικής σχέσης, ποιοι είναι οι εταίροι και το καθεξής. Και τι θα γίνει με το αδεοντολογικό κώδικα και σε σχέση με τις μειονότητες, ιδιαίτερα τους συγκάνους σε εκείνες τις χώρες κυρίως, όπου αυτό είναι ζήτημα, ζήτημα κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, ατομικό, προσωπικό υπό η αδίποτε τέτοια πτυχή για τι κοινότητες των Ρωμά, των Συγκάνων. Και αναμένουμε ότι και στα λειτουργικά προγράμματα θα ενταχθεί το ζήτημα των Ρωμά, των Συγκάνων και θα ε, εντάσσεται και θα παρουσιάζεται. Θέλω να μου δώσετε τη διασφάλιση αυτή από πλευρά ε, τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο στι διαβουλεύσει για την ε, εταιρική σχέση με εκείνε τι χώρε όπου αυτό το θέμα είναι σημαντικό, ότι αυτό θα ενταχθεί δηλαδή στην ημερήσια διάταξη ω θέμα τη Επιτροπή Ρέγγι και το ίδιο και για την απασχόληση. Δεν ξέρω πώ διαμορφώνουν, πώ θα αντιμετωπίζουν οι εθνικέ στρατηγικέ και πώ ε, συνοδεύει και εποπτεύει αυτέ τι Τυχέ των εθνικών στρατηγικών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό το πρίσμα μελλοντικού προπολογισμού. θέλουμε να συνεισφέρουμε ως Ευρωκοινοβούλιο να ληφθεί υπόψη το θέμα και να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση αυτή τη πρόκληση. Έχει υπόψη τη να διασφαλίσει αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επίπεδο κρατών μελών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Πράγματι αυτό που κάνουμε τώρα είναι να ευαισθητοποιήσουμε και του αρμόδιου υπαλλήλου ε, από πλευρά μα. Καταρτίζουμε δηλαδή τους ε, αρμόδιους υπαλλήλου που θα επομιστούν το θέμα διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη για αυτή την ε, υπόθεση. Στοχοθετημένε δράσει για τα θέματα των συγκάνων, για την θεσμοθέτηση και θεσμική διάσταση που πρέπει να εντάσσεται. Στοχοθετημένη κατάτηση και εκπαίδευση για την ε, ένταξη των Ρωμά των Τσιγκάνων σε μια ολοκληρωμένη πολιτική, κοινωνική πολιτική, συγκεκριμένα με τι ανάγκε κάθε χώρα και πώ όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτική από πλευρά μα. Αυτό κάνουμε. Και πράγματι ο λόγο για τον οποίο ε, παρίσταμε είναι ότι εμεί στην γενική μα διεύθυνση έχουμε ένα τμήμα αρμόδιο όπου εγκάρσει ε, επιλαμβάνονται των θεμάτων των συγκάνων και έχουμε την ευθύνη να ε, ερχόμαστε σε επικοινωνία και σε διασύνδεση με τους άλλους συναδέφους άλλων ε, τμήματων και υπηρεσιών ώστε τα θέματα των συγκάνων να είναι αλληλένδετα από πλευρά μα. Ε, θα εξετάσουμε λοιπόν όλα αυτά σε πολλέ πτυχέ, πολυσύνθετα, πολυδιάστατα, ώστε να συνδέονται, αλληλοσυνδέονται σε σχέση με τα έγγραφα που θα συνταχθούν και θα παραθούν από πλευρά μας αυτά τα θέματα δεν υπάρχει άλλο που να θέλει να ζητήσει τον λόγο για σχόλια. Σα ευχαριστούμε πολύ για αυτέ τι πληροφορίε. Από ό,τι γνωρίζουμε θα είσαστε σε για, είμαστε σε επαφή για οποιαδήποτε θέματα όσον αφορά για παράδειγμα την ακρόαση αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι ότι η επόμενη συνεδρίασή μα θα διεξαχθεί στι 19 Φεβρουαρίου. Με αυτή την πληροφορία λίγη συνεδρίασή μα ε, και τερματίζονται οι εργασίε μα, σα ευχαριστώ. Γεια σας.